Καλή σας μέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Παρακαλώ καθίστε για να ξεκινήσουμε. Θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας με το σημείο 9. Πρόγραμμα κατοχώρησης ταξιδιωτών. Η συγητής είναι ο συνάδελφος Γιώαν Ένσιου. Θα έχουμε κοινή συζήτηση. Θα συζητήσουμε δηλαδή μαζί το 9 και το 10 για το σύστημα εισόδου-εξόδου για την καταχώρηση δεδομένων εισόδου και εξόδου των υπηκών τρίτων χωρών που διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγγήτρια για το θέμα αυτό είναι η κυρία Ρενάτε Σόμερ. Στόχος είναι να εξετάσουμε τα, τα έγγραφα εργασία και προτείνω να ακούσουμε πρώτα τους δύο εισηγητές. Να ακούσουμε κατόπιν τον κύριο Πίξπαν που ε, ε, είναι εκπρόσωπος του ε, Ευρωπαίου Επόπτη για τα προσωπικά δεδομένα. και της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 οι οποίοι θα μας ε, δώσουν τις γνωμοδοτήσεις τους και μετά θα ακούσουμε την ε, Κομισιόν, το Συμβούλιο και τους ε, Ευρωβουλευτές. Παρακαλώ λοιπόν. Να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Ένσιου και μετά την κυρία Σόμερ. Yes, Mr. Would like to go first, Sommer?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 Η πρόταση συστήματος εισόδου-εξόδου ε, αποτελεί μέρος ε, του πακέτου για τα FEE e σύνορα. Οι ε, πήκοοι τρίτων χωρών γενικά μέσα σε έξι μήνες σε ένα διάστημα έξι μπορούν να μείνουν μέχρι τρεις μήνες στην περιοχή Σέγγεν. Αυτή τη στιγμή αυτό ελέγχεται με σφραγίδες στα διαβατήρια. Μέχρι στιγμής δηλαδή δεν υπάρχει ηλεκτρονική καταχώρηση ε, του πότε ε, διέθετε κανείς από την ε, ζώνη Σέγγεν. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει επιγόντως, δεδομένου ιδιαίτερως ότι προβλέπονται όλο και περισσότερες απελευθερώσεις θεωρήσεων για υπηκόους τρίτων χωρών. Με την πρόταση αυτή λοιπόν τι θέλουμε να πετύχουμε. Ε, οι σφαγίδες στα διαβατήρια είναι κάτι χρονοβόρο και δύσκολο. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο ε, να ελέγξει κανείς 20 ε, σφαγίδες εάν κάποιος υπηκός τρίτων χωρών έχει περάσει 10 φορές από την ζώνη Σέγγεν. Οι σφαγίδες μπορούν να είναι πλαστές. Επιπλέον υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν έχουμε ενιαίο, εν, εν, ενιαία καταχώρηση ε, εισόδου και εξόδου από τη ζώνη Σέγγεν, ε, οπότε δεν μπορούμε να δούμε ε, εάν κάποιος έχει μείνει παραπάνω από ό,τι του επιτρέπεται. Για υπηκό τρίτων χωρών, των οποίων τα, δεδομένα, τα βιομετρικά δεδομένα δεν υπάρχουν στο σύστημα VIS και των οποίων έχουν καταστραφεί τα διαβατήρια, δεν μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτότητά τους. Ε, οι χώρες του Σέγγεν, 13 χώρες έχουν ε, κάποια δικά τους ε, συστήματα, αλλά δεν είναι δυνατόν να ελέγξει κανείς αξιόπιστα την έξοδο από τη ζώνη Σέγγεν υπηκών τρίτων χωρών. Γι' αυτό θα πρέπει τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα να τους προσαρμόσουμε στις τεχνικές δυνατότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Χρειαζόμαστε σύγχρονα και αποτελεσματικά όργανα για έλεγχο και εφαρμογή των κανόνων. Οι έλεγχοι θα πρέπει να απλοποιηθούν όσο γίνεται και να αυτοματοποιηθούν. Κάτι το οποίο θα ωφελήσει όχι μόνο τους ταξιδιώτες, αλλά θα βοηθήσει και εμάς να ελέγξουμε την ε, λάθρο μετανάστευση και με το ε, σχετικό σύστημα θα μπορέσουμε την ε, μελλοντική πολιτική για τις θεωρήσεις ε, να την ε, στοχεύσουμε περισσότερο στα βασικά θέματα και τα βιοματρικά δεδομένα υπηκών τρίτων χωρών που εισέρχονται στη ζώνη Σέγγεν θα καταχωρούνται και όχι μόνο αυτά των υπηκών για τους οποίους υπάρχει υποχρέωση θεώρησης. Το σύστημα λοιπόν ε, καταχώρησης και αποθήκευσης ε, των ε, πληροφοριών αυτών θα δίνει και ειδοποίηση όταν έχει εκπνεύσει το χρονικό διάστημα μόνιμης παραμονής. Ε, επίσης ε, θα υπάρχει φάκελος ε, ατομικός για κάθε ταξιδιώτη όπου θα υπάρχουν προσωπικά δεδομένα όπως είναι όνομα, είδος και αριθμός ταξιδιωτικού εγγράφου και ενδεχομένως αριθμός της θεώρησης. Για τους ανθρώπους που δεν έχουν, για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση θεώρησης, δηλαδή τα άτομα των οποίων τα δαχτυλικά αποτυπώματα δεν υπάρχουν στο VIS και που στο παρελθόν δεν συμπεριλαμβάνονταν, θα υπάρχουν υπάρχει προσωπικό φάκελο σε μέρα χτυλικά αποτυπώματα. Ε, για κάθε μετακίνηση των ανθρώπων αυτών ε, θα ε, αναφέρεται ο τόπος και η ώρα εισόδου στο Σέγγεν, στην ζώνη Σέγγεν. Η πρόσβαση προς το σύστημα αυτό Οι αρχές θα μπορούν να ελέγξουν τις ε, αιτήσει ε, και θα ε, ελέγχεται η ταυτότητα των, ε, ταξιδετών, τρίτων χωρών και θα διαπιστώνεται εάν πληρώνουν τις προϋποθέσεις για παραμονή. Οι συνολικές αρχές και οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να έχουν πρόσβαση ε, με στόχο την ταυτοποίηση ατόμων και για τους ελέγχους των προϋποθέσεων για την παραμονή στην ζώνη Σέγγεν θα ισχύει η γενική απαγόρευση διαβίβασης δεδομένων από το σύστημα αυτό σε τρίτες χώρες ε, και εξαιρέσεις ε, θα υπάρχουν μόνο σε πολύ συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις. Όσον αφορά λοιπόν την αναγκαιότητα του συστήματος αυτό. Έχουμε ακούσει τη γνωμοδότηση της ε, ομάδας ε, του άρθρου 29. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο ένα τέτοιο σύστημα. Ε, μόνο όμως αν εκμεταλλευτούμε όλες του τις δυνατότητες και δημιουργήσουμε έτσι προστιθέμενη αξία στην ευρωπαϊκή πολιτική θεωρήσεων. Το σύστημα αυτό είναι αρκετά ακριβό και θα πρόκειται για μια πολύ μεγάλη βάση δεδομένων. Ε, ειδικό θέμα είναι η χρήση της βάσης δεδομένων ε, για την ε, δίωξη εγκλημάτων. Πιστεύω ότι για τέτοιους στόχους θα πρέπει να χρησιμοποιείται η βάση δεδομένων αυτή και ότι ήδη πολλά κράτη-μέλη χρησιμοποιούνται αυτή τη δυνατότητα και έχουν συλλέξει πολύ καλές εμπειρίες. Ιδιαίτερα θέλουμε διασυνοριακά εγκλήματα όπως είναι η τρομοκρατία, το λαθρεμπόριο κλπ. Ε, να τα αντιμετωπίσουμε και το σύστημα καταχώρησης μπορεί να συμβάλλει σημαντικά σε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει λοιπόν να εκμεταλλευτούμε τη δυνατότητα αυτή. Η χρήση βιομετρικών δεδομένων είναι άλλο θέμα. Η η Κομισιόν λέει ότι η χρήση βιομετρικών ε, δεδομένων ε, και η ε, χρήση τους για δίωξη εγκλημάτων θα είναι πολύ χρήσιμη στην καταπολέμηση τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων και ε, τα δακτυλικά αποτυπώματα είναι αξιόπιστο και ταχύ μέσο για τον έλεγχο της ταυτότητας του υπόπτου. Μόνο τα βιομετρικά δεδομένα ε, επιτρέπουν ε, γρήγορη και αξιόπιστη ταυτοποίηση και με τα στοιχεία αυτά θα αποδείξει την αξία του το σύστημα αυτό και είμαι πεπισμένη ότι αν ε, συλλέγουμε βιομετρικά δεδομένα επικών τρίτων ε, χωριών, ε, αυτό θα συμβάλλει σημαντικά σε μείωση της λαθρομετανάστευσης, διότι θα είναι δυνατή η ταυτοποίηση οποιοδήποτε επικό τρίτης χώρας που βρίσκεται στην, στην περιοχή μας η Κομισιόν στην πρότασή της ε, ήθελε ένα σύστημα το οποίο βασίζεται σε token. Αυτό υπάρχει στο άρθρο 27 θα πρέπει να υπάρχει τσιπάκι με ε, αριθμό ταυτοποίησης ε, που θα συγκρίνεται με ε, τα δεδομένα στη βάση. Αυτό ωραίο ακούγεται, αλλά νομίζω ότι είναι περιττό και απλά θα επιφέρει περιττό κόστος καθώς και τον κίνδυνο απώλειας και παραποίησης πιο χρήσιμο θα είναι να χρησιμοποιήσουμε το ηλεκτρονικό διαβατήριο. Το πρότυπο, ε, το, ε, το πρότυπο αυτό διαβατήριο το οποίο ε, ε, χρησιμοποιείται όλο και σε περισσότερες χώρες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως token. Και Και έτσι μπορούμε να αποφύγουμε και το επιπλέον κόστος που θα έχουμε αν έχουμε μια κάρτα με τσιπάκι. Ε, τα δαχτυλικά αποτυπώματα ως μοναδικό ε, σύστημα ταυτοποίησης ε, θα πρέπει, μέχρι στιγμής θα πρέπει να συμπληρωθεί από φωτογραφία. Ε, το token ε, θα είναι ιδιαίτερο ακριβό σύστημα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν σύστημα βασισμένο ε, στα βιομετρικά δεδομένα και έχουν απολύτω θετικέ εμπειρίε Γιατί λοιπόν να μην μάθουμε κι εμείς από τι εμπειρίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν νομίζω ότι σε εποχές λιτότητας θα είναι ότι θα είναι καλό να δώσουμε πολλά χρήματα για συστήματα για τα οποία ήδη από την αρχή υπάρχει αμφιβολία εάν θα λειτουργήσουν επιτυχώς τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν άλλα συστήματα που λειτουργούν ε, πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Με χαρά σας παρουσιάζω αυτό το έγγραφο εργασίας το οποίο παρουσιάζει συνοπτικά την πρόταση, ιδιαίτερα συνοπτικά, αλλά θέτει νομίζω κάποιες πολιτικές ερωτήσεις. Βασικός στόχος του RTP είναι να διευκολυνθεί το πέρασμα σε πολίτες των τρίτων χωρών των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που έχουν εμποδιστεί πριν φτάσουν στα σύνορα. Between travelers from third countries. Το RTP λοιπόν travel flows and expect... Βασικός στόχος είναι να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ταξιδιώτες αυτοί στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών είναι η σωστή διαδικασία. Κάθε πολίτης άνω των 12 ετών από τρίτη χώρα μπορεί μέσω του RTP να κάνει μία αίτηση σε οποιοδήποτε ε, προξενείο χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να παρουσιάσει ένα μηχανικά αναγνώσιμο ταξιδιωτικό έγγραφο και θα πρέπει να πληρώσει επίσης ε, ένα παράβολο 20 ευρώ. Το θέμα το οποίο πτήθεται προς συζήτηση νομίζω είναι μία σειρά ερωτήσεων που χρήζουν απαντήσεων. Πρώτον, καταλληλότητα του συστήματος ως έχει. Θα πρέπει να γνωρίζουμε εάν πράγματι χρειαζόμαστε το ATP και αν υπάρχουν εναλλακτικές σε αυτό λύσεις. Τον Μάρτιο του 2009 το Κοινοβούλιο υποστήριξε καταρχάς την ιδέα δημιουργίας του RTP για τους πολίτες τρίτων χωρών. Υποστήριξε λοιπόν την ιδέα του RTP, αλλά θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να σκεφτούν από το αν θα μπορούσαν να υπάρξουν και διαφορετικές λύσεις για τους εξωτερικούς τελωνιακούς ελέγχους. Υπάρχει δυνατότητα να αυξηθούν ε, οι αριθμοί των ανθρώπων που διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα. Τα τελευταία τρία χρόνια δεν έχει υπάρξει μια τέτοια αύξηση. θεωρείται επίσης από το, ε, από το σύστημα το οποίο έδωσε αν θέλετε την δυνατότητα δημιουργίας του RTP ότι η πίεση σε όλες τις χώρες ε, της ζώνης Σέγγεν με τον ίδιο τρόπο, ότι υπάρχει η ίδια πίεση σε όλες αυτές τις χώρες, κάτι το οποίο δεν είναι αλήθεια. Ο μεγάλος αριθμός των περασμάτων των εξωτερικών συνόρων γίνονται βασικά από ε, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολίτες τρίτων χωρών που έχουν όμως την δυνατότητα ελεύθερης διακίνησης νομίμως. Υπάρχουν πολίτες από τρίτες χώρες που έχουν νόμιμα δικαιώματα σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα. Έχουν επίσης την δυνατότητα σαν παράδειγμα να φέρουν τα πρόσωπα της οικογένειάς τους. Μια άλλη ιδέα, πέρα από τα αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου, είναι να προβλέπονται δειγματοληπτικά ε, τέτοια συστήματα ελέγχου για αυτούς ε, οι οποίοι κατέχουν θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων. Ε, since the criteria, criteria for the issuing an MED are quasi the same as for the, for the RTP. Τα κριτήρια λοιπόν και για τα υπόλοιπα συστήματα θα πρέπει να είναι τα ίδια με τα κριτήρια που οδήγησαν στο RTP. Θα πρέπει να αποφύγουμε με αυτόν τον τρόπο τις επικαλύψεις με τα ισχύοντα συστήματα όπως το PIS. Η αυτόματη ή αυτόματη έλεγχη ε, στα εξωτερικά σύνορα, ιδιαίτερα και στους αερολιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βέβαια κατά πρώτον, θα είναι κάτι το οποίο θα μειώσει το χρόνο αναμονής. Ιδιαίτερα στα αεροδρόμια τα οποία έχουν υψηλή κίνηση. Λόγω και της οικονομικής κατάστασης ορισμένες χώρες μέλη έχουν προβλήματα συντήρησης των δημόσιων συστημάτων ελέγχου και γι' αυτό τίθεται εδώ το θέμα της σωστής εφαρμογής, δυνατότητας εφαρμογής του RTP. Μήπως θα πρέπει να δοθεί ε, βάρος και στις ε, δημοσιονομικές συνέπειες της πρότασης. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέγει ότι 585 εκατομμύρια ευρώ είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη του συστήματος αυτού. Όμως το συνολικό κόστος και σε εθνικό επίπεδο και σε κοινοτικό επίπεδο στα πλαίσια των υπολογισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται σε 712 ε, εκατομμύρια. Έχουμε λοιπόν μια διαφορά 125 εκατομμυρίων ευρώ. Και συνολικά τα ποσά θα ξεπεράσουν το 1 δις. όπως ακριβώς περιλαμβάνονται στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναμένουμε λοιπόν διευκρινήσεις σε σχέση και με το λειτουργικό κόστος των συγκεκριμένων προτάσεων και των δημοσιονομικών επιπτώσεων που θα προκαλέσει στα κράτη-μέλη εποχή μάλιστα δημοσιονομικής πίεσης πολύ σοβαρής. Το 1 δις 350 εκατομμύρια για την ανάπτυξη των λεγόμενων εφιών συνόρων είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προωθηθεί αλλά με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και πιθανές εναλλακτικές λύσεις. Ο υπολογισμός των εσόδων που υπολογίζεται ότι θα ε, δημιουργηθούν από την εφαρμογή του συστήματος RTP μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα ακριβής. Η Επιτροπή θεωρεί ότι 5 εκατομμύρια εγγραφές στο σύστημα RTP θα γίνονται σε ετήσια βάση. Όμως αυτό είναι αμφισβητήσιμο αν λάβουμε υπόψη μας το ότι το σύνολο των συμμετεχόντων στα αντίστοιχα ισχύοντα συστήματα στις χώρες οι οποίες έχουν ε, ε, αερολιμένες με πάρα πολύ μεγάλη κίνηση ε, δεν δικαιολογούν τους υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 45.000 στην Γερμανία, 48.000 στην Ολλανδία, 500, 500 ε, μόνο αιτήσει συμμετοχή στο Ιρκούτσκ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι το σύστημα RTP είναι τμήμα ενός συνολικότερου πακέτου. Στην πρώτη φάση μόνο με αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν σε συστήματα αντίστοιχα τα οποία είναι ενισχύ θα μπορούν να πάρουν μέρος. Έτσι όμως ε, θα διευκολυθούν σίγουρα οι διαδικασίες και θα καταργηθεί και η σφραγίδα στο αδιαβατήριο. Ένα RTP ε, θα μπορεί να ξεκινήσει σχετικά εύκολα χωρίς να ληφθούν υπόψη τα ισχύοντα συστήματα, κάτι όμως ε, το οποίο για μία μακρά περίοδο θα απαιτήσει την χρήση επίσης συνοριοφυλάκων ή τελωνοφυλάκων οι οποίοι θα πρέπει να σφραγίζουν τα ταξιδιωτικά έγγραφα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 στον κύριο Χίτμαντ, που είναι εκπρόσωπος ε, του, Ευρωπαϊ... Ε, του Ευρωπαίου Πόπτη για τα προσωπικά δεδομένα. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μας δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσουμε την ε, γνώμη μας τη 18 Ιουλίου να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του κ. Χάστιν και κ. Κουρτακέλη που δεν ε, βρίσκονται σε θέση να παρευρεθούν στη σημερινή συνεδρίαση. Θα πρέπει να αρκεστείτε σε μένα. Θα επικεντρωθώ στο σύστημα εισόδου-εξόδου ε, καθότι ε, εδώ προκύπτουν τα πιο θεμελιώδη ερωτήματα όσον αφορά την προστασία του ιδιωτικού βίου και την προστασία των δεδομένων. Ε, στο πρόγραμμα καταχώρησης ταξιδιωτών θα αναφερθώ σύντομα στο τέλος της παρέμβασής μου. Ε, εξετάσαμε τα έγγραφα που ετοίμασαν οι ε, εισηγητές και νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο να επικεντρωθούμε στα δύο θέματα που έθιξε η κυρία Σόμερ, την αναγκαιότητα δηλαδή και τις ρυθμίσεις του συστήματος συστήματος. Στη γνωμοδότησή μας παρέχουμε ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση της ε, ε, ε, συμβατότητας ενός τέτοιου μεγάλου συστήματος όπως είναι το σύστημα καταχώρησης εισόδου-εξόδου με τον χαρτί θεμελιωτών δικαιωμάτων. Υπάρχει λοιπόν το θέμα της ε, χρήσης δύο ε, κατοφλίων ε, για τον έλεγχο αυτών. Το ένα είναι ο σεβασμός του οικογενειακού βίου. Ένα σύστημα εισόδου-εξόδου παραβιάζει αυτό το δικαίωμα και θα πρέπει να εξεταστεί αν είναι αιτιολογημένη μια τέτοια. Το άρθρο λοιπόν αυτό είναι το πρώτο κατόφλι το οποίο θα πρέπει να ε, σχετιστεί με την απάντηση που θα δοθεί στο ερώτημα της ε, ε, κυρίας Σόμερ την αναγκαιότητα του συστήματος. Κατόπιν έχουμε το άρθρο 8, το οποίο επιτρέπει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εφόσον πληρούνται κάποια βασικά κριτήρια. Το άρθρο 8 λοιπόν καθορίζει τους κανόνες για την επεξεργασία δεδομένων. Το ερώτημα λοιπόν εδώ είναι το σύστημα καταχώρηση του εξόδου πληρεί τις βασικές αυτές προϋποθέσεις, με άλλα λόγια το άρθρο 8 θα πρέπει να απαντήσει στο ερώτημα της κυρίας Σόμερ εάν οι, ρυθμίσεις, οι επιμέρους ρυθμίσεις της πρότασης αυτής ε, ε, συνάδουν με τον ε, χάρτη προστασίας δεδομένων. Πιστεύουμε λοιπόν ότι ένα ολοκληρωμένο σύστημα όπως το σύστημα, ότι για ένα τέτοιο σύστημα καταχώρησης εισόδου-εξόδου είναι χρήσιμο να εξετάσουμε τα δύο αυτά κατόφλια, να κάνουμε αυτή τη διπλή δοκιμή. Και με βάση τα ερωτήματα αυτά υπάρχουν βασικές αμφιβολίες σχετικά με την αναγκαιότητα του συστήματος και σε, επιστολή μας επικρίνουμε και τις ε, ρυθμίσεις της πρότασης. Η βασική μας ε, όμως συμβουλή είναι να χρησιμοποιηθεί αυτό το πλαίσιο αξιολόγηση Ω ε, ως μέρος της ε, διαδικασίας ε, λήψης αποφάσεων με την οποία δεν θέλουμε να παρέμβουμε. Το σύστημα αυτό είναι ολοκληρωμένο. Θα πρέπει λοιπόν να βασιστεί η δημιουργία του σε διάφορου τέτοιου συλλογισμού. Κατά τη γνώμη μα, αυτό προβλέπει και το σύστημα τη Στοκχόλμη. Νέα συστήματα θα πρέπει να αναπτύσσονται μόνα όταν διαπιστώνεται ότι τα υπάρχοντα δεν αρκούν. Σημειώσαμε ότι ε, από την έναρξη του προγράμματος της ε, η Κομισιόν διστάζει πολύ να εισάγει νέα συστήματα. Γι' αυτό ακριβώς ε, μας κάνει εντύπωση που προτείνεται το σύστημα καταχώρησης οδεξόδου ε, τη στιγμή που ήδη υπάρχουν μεγάλα συστήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που σχετίζονται με, το, με τους συναριακούς ελέγχους. Επιπλέον ε, τα δύο ε, βασικά ε, συστήματα δεν έχουν τεθεί πλήρως σε ισχύ και φυσικά δεν έχουν αξιολογηθεί επίσης το ΒΙΣ και το ΣΥΣ2 τέθηκαν σε ισχύ πολύ πρόσφατα και με βάση αυτά θα πρέπει να εξεταστεί το σύστημα καταχώρησης ξόδου. Να προχωρήσω τώρα στην αναγκαιότητά του και, τον, και το άρθρο 7 του Χάρτη ε, Θεμελιωτών Δικαιωμάτων. Δεν ε, συμμεριζόμαστε όλες τις συστάσεις ε, του εισηγητού. Ε, διαφωνούμε και να είμαι ακριβής. Ε, εξετάσαμε την συμβατότητα με το άρθρο 7 του Χάρτη ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, και εξετάσαμε τον στόχο του συστήματος αυτού. Ο βασικός στόχος του συστήματος αυτού είναι να καταπολεμήσει το φαινόμενο να παραμένει ένας ταξιδιώτης μετά την... αφού, αφού το εκμεύσει το διάστημα όπου έχει δικαίωμα να παραμείνει στην Ένωση. Ένα τέτοιο σύστημα, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να καταπολεμήσει το φαινόμενο αυτό, θα πρέπει πρώτα να αναπτύξει μια ε, συνεκτική πολιτική και κατόπιν ε, το σύστημα αυτό να αποτελέσει μέσο της ε, πολιτικής αυτής, ε, όπως ε, το σύστημα πληροφόρησης Schengen ήταν ένα απαραίτητο εργαλείο όταν δημιουργήθηκε ο χώρος Schengen. Αλλά αυτή τη στιγμή το σύστημα αυτό δημιουργείται ως ανεξάρτητο σύστημα, χωρίς την απαραίτητη νομοθεσία και αναρωτιόμαστε αν αυτή είναι η σωστή σειρά να γίνουν τα πράγματα. Επίσης, όσον αφορά την συλλογή δεδομένων ως ξεχωριστό στόχο που αναφέρεται στην πρόταση αυτή, θεωρούμε ότι αυτό είναι ένας επιπλέον στόχος και όχι ο βασικός στόχος του συστήματο καταχώρηση καταχώρησης εισόδου-εξόδου. Καταλαβαίνουμε ότι χρειάζονται σωστέ στατιστικές ε, για να καταπολεμηθεί το φαινόμενο ε, της ε, παραμονής όταν δεν έχει πια κανείς δικαίωμα να παραμείνει, αλλά δεν αρκεί το να αποθηκεύσουμε και να καταχωρήσουμε ανώνυμα δεδομένα για κάτι τέτοιο. Και τέλος αναφέρθηκε η ανάγκη για εξυγχρονισμό των συνοριακών ελέγχων. Δεν είμαστε, κατά κάτι, δεν είμαστε ε, αντίθετοι με κάτι τέτοιο, αλλά ε, προκύπτει το ερώτημα αν ε, αυτό θα πρέπει να γίνει με μια τεράστια βάση δεδομένων. Να προχωρήσω γρήγορα τώρα στο άρθρο 8. Η υπηρεσία μας επίσης εξέτασε την, τη συμβατότητα με τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εξετάσαμε δηλαδή τις ε, μέρου ρυθμίσει ε, τη πρόταση, ε, όπως αναφέρονται στην έκθεση της κυρίας Σόμερ. Δεν θα σας επαναλάβω αναλυτικά το, το, το τεστ αξιολόγηση. θα αναφέρω μόνο τα πιο βασικά στοιχεία. Καταρχήν, περιορισμός του στόχου θα ε, απαιτήσει οι στόχοι της πρότασης να γίνουν πιο συγκεκριμένοι. Επίσης, το σύστημα δεν θα πρέπει να βασίζεται σε πιθανή πρόσβαση για την επιβολή του ε, νόμου. Για, το, για τα όργανα επιβολής του νόμου. Θα πρέπει το σύστημα αυτό να δομηθεί με τρόπο ώστε να προστατεύει τον ιδιωτικό βίο. Το άρθρο 8 του χάρτη δεδομένων, ε, του Δικαιωμάτων επίσης Ε, αναφέρει ότι δεν θα πρέπει να είναι ε, υπερβολικά τα μέτρα. Η πρόταση αυτή δεν είναι υπερβολικό πράγματι όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Ε, ωστόσο, προτείνουμε να είμαστε πιο αυστηροί όσον αφορά τα βιομετρικά δεδομένα και θα θέλαμε να περιοριστούμε σε δύο ή τέσσερα δακτυλικά αποτυπώματα και όχι ε, δέκα όπως προτείνεται τώρα για το πρόγραμμα καταχώρησης ταξιδιωτών. Ε, να επανέλθω ε, σύντομα στο σύστημα καταχώρησης εισόδου-εξόδου από πλευράς της προστασίας των δεδομένων χωρίς να αναφερθούμε καθόλου στους συλλογισμούς του κυρίου Ένσου Πιστεύουμε ότι η πρόταση αυτή είναι λιγότερο προβληματική, είναι ε, προαιρετικό το σύστημα και θα διευκολύνει την, ε, τους συνοριακούς ελέγχους ε, για τους ανθρώπους που ταξιδεύουν συχνά. Αλλά το βασικό μας μέλημα είναι το σύστημα αυτό να παραμείνει προ, προαιρετικό. Να μην είναι αναγκαστικό και να ε, διασφαλίσετε ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις ε, για κάποιον ε, που αρνείται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα αυτό. Δύο τελικές παρατηρήσεις το πρόγραμμα εποπτείας που προβλέπεται είναι αυτό που ισχύει αυτή τη στιγμή για τη Eurodac, για το SIS και για το VIS. εποπτεύεται από την Ιουλίσα e και υπάρχει στενή συνεργασία με τις εθνικές αρχές. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια σοφή επιλογή η οποία ταιριάζει απόλυτα με την ε, δημιουργία του χώρου ε, ελευθερίας ε, ειρήνης και δικαιοσύνης ασφαλείας και δικαιοσύνης. όσον αφορά τις τεχνικές συστάσεις που έχουμε υποβάλει, προτείνουμε στην Επιτροπή σας να τις εξετάσετε. Ε, ιδιαίτερα εκεί που μιλάμε για ε, συνέχεια και συνέπεια στην εφαρμογή των κανόνων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Και τώρα να ακούσουμε τον εκπρόσωπο της ομάδας του άρθρου 29, της ομάδας εργασία του άρθρου 29, τον κύριο Μπέν. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Να σα ευχαριστήσω εκ μέρου τη ομάδα εργασία που μα δίνετε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε τη δική μα την ε, τοποθέτησή σε σχέση με το θέμα. όπως και η DPS, εγώ θα μιλήσω για το σύστημα εισόδου-εξόδου, γιατί είναι το πλέον ενδιαφέρον σε σχέση με το έργο μας. Τι λέμε στην δική μας τη γνωμοδότηση, την ανάγκη να υπάρχει ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, όπως και το γεγονός ότι η αναχέτηση της λαθρομετανάστευσης είναι ένας από τους βασικότερους βεβαίω, αλλά ολοκληρώνουμε ζητώντας να γίνει πιο αποτελεσματικό το σύστημα εισόδου-εξόδου, λέγοντας ότι οι ανάγκες και η αναλογικότητα είναι κριτήρια τα οποία δεν έχουν γίνει αρκετά σεβαστά. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να σας εξηγήσω γιατί καταλήξαμε σε αυτό το συμπέρασμα. Η Επιτροπή εντοπίζει διαφορετικούς λόγους για τη δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος εισόδου-εξόδου για να αντιμετωπιστεί η έλευση μεταναστών στην ε, Ευρώπη για την παράνομη μετανάστευση αλλά η ομάδα εργασίας θεωρούσε ότι αυτό δεν είναι αρκετά αποτελεσματικό και πιστικό για τους εξής τρεις λόγους. Πρώτον, το σύστημα αυτό μπορεί να είναι λειτουργικό. Εδώ ήδη έχουμε κάποιες πρώτες αμφιβολίες. Το σύστημα εν γέννη θα είχε νόημα εάν χρησιμοποιείτο ε, και επέτρεπε να θεωρήσουμε ότι οποιαδήποτε είσοδος και έξοδος ε, παράνομων ή άτυπων μεταναστών από τα εξωτερικά σύνορα θα καταγράφονται σωστά. Όμως είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει ένα τέτοιο σύστημα το οποίο θα προβλέπει την καταγραφή ειδικά της εξόδου στις Ηνωμένε Πολιτείες δεν έχει καταφέρει το αρμόδιο Υπουργείο να δημιουργήσει ένα τέτοιο σύστημα. Εάν σκεφτούμε και τη γεωγραφική κατανομή της Ευρώπης, το πόσο εκτεταμένα είναι τα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορά μας, το πόσα πούλμαν, λεωφορεία, τρένα, ε, ferry boat ε, κυκλοφορούν μεταξύ Ευρώπης και των υπόλοιπων υπηρών Βορείου, Αφρικής και Ασίας είναι πολύ δύσκολο να δημιουργηθεί ένα τέτοιο σύστημα. Θα πρέπει να σκεφτούμε επιπλέον τις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν. Και δεν είναι μόνο τα στατιστικά δεδομένα, το κατά πόσον θα ήταν ορθά ή όχι αυτά που θα συλλέγαμε. Αλλά είναι και το θέμα των ε, λανθασμένων, των εσφαλμένων ειδοποίησεων ή των ε, λαθανσμένων καταγραφών στοιχείων. Εάν υποθέταμε λοιπόν ότι έχουμε πιστεί ως Ευρωπαϊκής Ένωση να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο σύστημα και απαντούσαμε και σε αυτό το πρώτο σημείο που έχω γύρει την αμφιβολία αυτή, αν απαντούσαμε καταφατικά, θα πρέπει να σκεφτούμε το εξή. Μπορεί το σύστημα αυτό να συμβάλλει σε κάτι στη διαχείριση των συνόρων. Το σύστημα αυτό λοιπόν θα μπορούσε ενδεχομένω να καταγράφει αυτού που παραμένουν περισσότερο χρόνο στην επικράτεια τη Ευρώπη, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα. Όπω του λόγου για του οποίου έχουν παραμείνει αυτοί στην επικράτεια, έπειτα τι γίνεται με αυτού που ε, φτάνουν στην Ευρώπη αλλά δεν φεύγουν με, για θεμετού λόγου για νόμιμους λόγους και έπειτα για το κατά πόσον θα υπάρχει η ανάλογη ανείχνευση. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να σκεφτούμε ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε παλιότερη ανακοίνωσή της εξηγούσε ότι το μείζον πρόβλημα είναι η επιστροφή ως προ την υλοποίηση. Εδώ δεν μπορεί να προσφέρει και πολλά το σύστημα εισόδου-εξόδου. Έτσι, Φτάνω στην τρίτη ε, βασική μου ε, αμφιβολία, στο βασικό μου ενδιασμό. Ποια θα είναι η συνεισφορά του συστήματος εισόδου-εξόδου προκειμένου να εντοπιστούν οι παρανόμως διαμένοντες στην επικράτεια της Ευρώπης. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί αν είχαμε τα ανάλογα βιομετρικά δεδομένα. Όμως σκεφτείτε το εξής. Εάν δημιουργηθεί αυτό το σύστημα θα πρέπει να βασιστεί σε όσα ήδη είχαμε στα χέρια μας, συγκεκριμένα το SIS2 και το BIS2, που περιλαμβάνουν βιομετρικά δεδομένα. Άρα το σύστημα εισόδου-εξόδου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως προς την ταυτοποίηση μόνον για τους επικός των χωρών αυτών όπου υπάρχει συμφωνία διευκόλυνση διευκόλυνσης θεωρήσεων. Άρσης μάλλον θεωρήσεων. Δηλαδή χώρες που εν γέννη γίνονται αντιληπτές ως χώρες που δεν παρουσιάζουν κίνδυνο λαθρομετανάστευσης. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε τις αμφιβολίες μας. Ε, αμφισβητούμε το κατά πόσο θα είναι αποτελεσματικό ένα τέτοιο σύστημα εισόδου-εξόδου. Να αναφέρω και άλλα τρία ζητήματα. Πρώτον, στατιστικά στοιχεία. Εάν η συνεισφορά για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης ή της άτυπης μετανάστευσης περιοριστεί τότε δεν είναι δικαιολογημένο να δημιουργούμε μια τεράστια βάση δεδομένων με όλα αυτά τα στατιστικά αποτελέσματα. Αλλά ακόμη και αν ήταν καλά τα στατιστικά στοιχεία θα μπορούσαν να αμφισβητηθούν. Διότι όσοι ε, φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και περνούν τα σύνορα παρανόμως δεν θα περιλαμβάνονται σε αυτές τις στατιστικές. Το δεύτερο ζήτημα είναι το κόστος. Αυτό δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με την προστασία των δεδομένων. Αλλά θεωρήσαμε ότι και αυτό είναι σημαντικό να ακουστεί Αναφέρθηκε και προηγουμένω στη συζήτησή σα αυτό η πρόσβαση στι ε, αρχέ καταστολής και για σκοπούς που εξυπηρετούν αυτές στα δεδομένα. Αυτό πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη προκειμένου να λάβουμε τη σωστή απόφαση. Εάν σκεφτούμε όλες αυτές τις παρατηρήσεις, νομίζω ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε και να τηρήσουμε μια πιο κριτική οπτική γωνία ως προς το σύστημα αυτό. Τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει και επαναλαμβάνει διαρκώς πόσο μεγάλη είναι το μεγάλο το ενδιαφέρον τη για την προστασία των δεδομένων, ένα τέτοιο σύστημα θα ήταν λανθασμένο μήνυμα προς τα έξω, πιστεύω. Αυτά είχα να πω για το EES, το σύστημα εισόδου-εξόδου, αλλά για να μην μακρηγορήσω, λίγα λόγια μόνον για το ε, σύστημα όπου ακούσαμε την κυρία Σόμερ το πρόγραμμα καταχώρησης ε, ταξιδιωτών για το οποίο ακούσαμε την κυρία Σόμερ να αναφέρει τις απόψεις της για το κατά πόσον θα χρειαζόταν εδώ μια βάση δεδομένων ή μήπως θα μπορούσαμε να βασιστούμε απλώς στα e-passes που ήδη χρησιμοποιούνται. Έχω και κάποια ακόμη σχόλια, αλλά επειδή δεν υπάρχει πάρα πολλοί χρόνος, προτιμώ να παραμένω σε αυτά. Ευχαριστώ. Ωραία. Ας συζητήσουμε λίγο τώρα. Ε, ας πάρουν το λόγο οι σκιώδεις εισηγητές. Ε, ο κύριος Ένσου, έτσι κι είναι σκιώδης στην έκθεση της κυρίας Σόμερ. Ακούσαμε λοιπόν και τα επιχειρήματα και των δύο. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο συμπληρωματικό σχόλιο για την έκθεση στην οποία είστε σκιώδης. Ε, αν όχι να ακούσουμε τους υπόλοιπους σκιώδης εισηγητές. Κοιτάξτε ας ακούσουμε τους υπόλοιπους συναδέλφους και στο τέλος της συζήτησης ίσως κάτι να πούμε. Thank you, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολλά θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά θα ξεκινήσω με κάποια γενικά σχόλια. Τα θέματα της προστασίας των δεδομένων τα αφήνω εκτός. Γιατί είναι κατανοητό στο Κοινοβούλιο ότι απαιτείται σωστή προστασία των ιδιωτικών δεδομένων και αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί σε άλλα επίπεδα, εν πάση περιπτώσει, με άλλους εισηγητές κτλ. Πάντως, αυτό το οποίο με ανησυχεί γύρω από το θέμα των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών είναι οι δυνατότητες, θα έλεγα, μη νόμιμων χρήσεων αυτών των στοιχείων. Δεν θα ήταν σωστό να πω ότι δεν θα πρέπει να βασίζεται ένα πρόγραμμα σε, ε, στα Windows σαν παράδειγμα και θα έπρεπε να βασίζεται στο Linux αλλά αυτό είναι κάτι το διαφορετικό βέβαια το οποίο δεν είμαι το σωστό όπως είπα πρόσωπο για να το προτείνω. What kind of um, amounts we are going to speak about in the future? If you look at what's going on in the world αν δείτε το τι συμβαίνει στον κόσμο σήμερα θα δείτε ότι το 1 τρίτο του πληθυσμού αυτή τη στιγμή μετακινείται. Οι περισσότεροι βέβαια στο εσωτερικό των χωρών τους. Αλλά δεν θα πρέπει να θεωρήσετε ότι τα πράγματα είναι ρόδινα και ότι θα εξακολουθήσουν να είναι ρόδινα στο μέλλον με λίγους γενικά ανθρώπους οι οποίοι να μετακινούνται. Αντίθετα βλέπουμε ότι από όλα τα στοιχεία και των Ηνωμένων Εθνών και της ΥΠΑ ΕΕ της Αυμοστίας για τους πρόσφυγες ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι μετακινούνται. Και αυτό θα μεγεθυνθεί σαν φαινόμενο και στο μέλλον και επίσης θα είναι κάτι το οποίο θα χαρακτηρίζει και τις λεγόμενες νόμιμες μετακινήσεις αλλά και αυτές οι οποίες είναι εκτός νομοθεσίας. Αυτό είναι χαρακτηριστικό του ανθρωπίνου είδους η μετακίνηση. Οι τεχνικές λύσεις δεν είναι κάτι που θα με απασχολήσει γιατί νομίζω ότι δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας νομίζω ότι θα βρούμε τεχνικές λύσεις αποτελεσματικές εφόσον προσπαθήσουμε. Δεν είναι όμως αυτό το θέμα, είναι εκτός αν θέλετε τη συζήτησή μας αν δούμε αυτούς οι οποίοι παραμένουν, τους παραμένοντες, θα δούμε ότι είναι δύσκολο να υπολογίσουμε πόσοι είναι και από ποιες χώρες προέρχονται. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα δύσκολο το να υπολογίσουμε πόσοι είναι αυτοί. και είναι και κάτι το οποίο θα δυσκολέψει τη συζήτηση. Είναι ενδιαφέρον φαινόμενο αυτοί οι οποίοι λοιπόν παραμένουν σε μια άλλη χώρα. Αλλά είναι δύσκολο να βρούμε από πού έρχονται και από κάποια στιγμή και μετά ποια είναι αυτή τη στιγμή όπου σταμάτησα, όπου παρέμειναν σε μια άλλη χώρα. Και αυτοί επίσης χρειάζονται μια κάποια προστασία διαφόρων μορφών και είναι στις δυνατότητές μας. για την έκθεση του κυρίου Έντσιου. Στα πλαίσια μιας δημοκρατικής διαδικασίας έχουμε μια απόφαση κοινοβουλευτική που λέει ότι απαιτείται ένα τέτοιο πρόγραμμα και θα πρέπει να εμείνουμε στην απόφαση αυτή μέχρι στιγμή που θα αποφασίσουμε κάτι το διαφορετικό. να μην ξεκινήσουμε μια συζήτηση τώρα για το αν έχουμε μια απόφαση. Αυτό είναι εκτός συζήτηση. Υπάρχει απόφαση του Κοινοβουλίου. Και ισχύει η απόφαση αυτή όσο υπάρχει. Δεν πρέπει να ε, αναζητούμε, ή μάλλον αν θέλουμε να αναζητούμε λύσεις για να αλλάξουμε την απόφαση αυτή, μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά πάντως η απόφαση αυτή στη φάση που είμαστε ισχύει. Η αναγκαιότητα του RTP είναι κυρίως να διευκολύνει και να επιταχύνει τις ε, μετακινήσεις και να διευκολύνει και τις εμπορικές συναλλαγές. Είναι θετικό αυτό. Έχουμε την πρόταση της Επιτροπής, δεν ξέρω αν θα πρέπει να αναζητήσουμε άλλες λύσεις, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε με ποιο τρόπο είναι καλή η πρότασή της. για τα πιο συγκεκριμένα στο έγγραφο Έντσιους. Αν θα πρέπει να διευκολύνουμε περισσότερο τις, ε, τις διαβάσεις ε, για αυτούς οι οποίοι έχουν το δικαίωμα ε, να περνούν από τα εξωτερικά σύνορα. Όχι δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι να διευκολύνουμε τις κινήσεις κατά πρώτον των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ το RTP αφορά τους πολίτες τρίτων χωρών. Τώρα, για το αν μπορούμε εμείς να μετροποποιήσουμε τον τελωνιακό κώδικα του, ε, του Schengen, έτσι ώστε να υπάρχουν αυτοματοποιημένοι έλεγχοι για αυτούς οι οποίοι έχουν θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων, τότε σε αυτή την περίπτωση κύριε Έντσου γιατί να μην γίνεται αυτό και από το RTP. Ακριβώς ε, τα ευφυή e e λεγόμενα σύνορα έχουν σαν στόχο να μην υπάρχουν διακρίσεις ανάμεσα στους πολίτες της Ένωσης και τους πολίτες των τρίτων χωρών και να μην υπάρχουν διακρίσεις ανάμεσα σε αυτούς που έχουν θεώρηση και σε αυτούς που δεν έχουν. Να μην δημιουργείται λοιπόν σύγχυση. Για να κλείσω λοιπόν αυτοί που έχουν ε, πολλαπλές ε, ε, μετακινήσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εν μέρη καλύπτονται από τις προτάσεις οι οποίες γίνονται και δεν είναι εύκολο να τους διευκολύνουμε ακόμα περισσότερο. Στα πλαίσια αυτής της συζήτησης ακούστηκε ότι το θέμα είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο τα αεροδρόμια και τους επιβάτες των αεροπορικών μεταφορών. Ε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι Ρώσοι που έρχονται στη Φιλανδία για πολλούς λόγους, νόμιμοι είναι όλοι σχεδόν, είναι τόσο ψηλός που δεν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό μόνο με αυτοματοποιημένες μεθόδους σε επίπεδο αερολιμένων. Τώρα έρχομαι στο κείμενο της κυρίας Ζώμεα. Θα ήθελα να μπορώ να μιλήσω γερμανικά, αλλά δεν είναι τόσο καλά τα γερμανικά μου ώστε να τα καταφέρω. Ε, Οπότε θα επανέλθω στα αγγλικά. I think that ε, Νομίζω ότι υπάρχει κάποια σύγχυση. Νομίζω ότι συμφωνούμε εν πολλής με την κυρία Ζώμα. Αλλά όπως είπα, δεν θα πρέπει να εξετάσουμε ιδιαίτερα και αποκλειστικά σχεδόν το θέμα αυτό των παραμενόντων. Together find some solutions on all the problems we have mentioned here. Now I've been speaking too long already, so thank you, Mr. Chair. Okay και Έκανε πρόταση ολόκληρη. Η... Η κυρία Κέλλερ, ευχαριστώ πολύ. Ε, με το πρόγραμμα εισόδου-εξόδου και λοιπά, θα δημιουργούσαμε την μεγαλύτερη βάση δεδομένων ε, και ε, δακτυλικών αποτυπωμάτων στον κόσμο, πράγμα προβληματικό ούτως ή άλλως. Ε, αν δεν γνωρίζουμε καν γιατί το κάνουμε, τότε έχουμε πραγματικά ένα μεγάλο πρόβλημα μπροστά μας. Με το σύστημα καταχώρησης εισόδου-εξόδου θέλουμε να διαπιστώσουμε πώς οι άνθρωποι παραμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την έκπνευση της θεωρησής τους ε, αλλά ε, εάν απλά θέλουμε να πετύχουμε καλές στατιστικές, ε, τότε συμφωνώ με τους εκπροσώπους του επόπτη προσωπικών δεδομένων. Δεν χρειαζόμαστε μια τόσο μεγάλη βάση δεδομένων για το θέμα αυτό. Και επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι δεν έχουμε καν ε, ε, κοινή πολιτική. Τι θέλουμε να κάνουμε με τους ανθρώπους αυτούς. Ε, έχουμε 26 διαφορετικές πολιτικές, διότι ρυθμίζεται διαφορετικά το ζήτημα αυτό στις διάφορες χώρες. Και τη στιγμή που δεν έχουμε κοινή πολιτική, νομίζω ότι έχει πολύ λίγο νόημα να έχουμε κοινή βάση δεδομένων και κατόπιν έχουμε και το κόστος. Ε, η ε, Κομισιόν υπολογίζει ήδη πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Ε, γνωρίζουμε όμως από άλλα μεγάλα συστήματα τέτοια ότι το κόστος αυτό μπορεί να αυξηθεί δραματικά και στις Ηνωμένε Πολιτείες το ελεγκτικό συνέδριο σταμάτησε το πρόγραμμα εισόδου-εξόδου. Αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, έχουν μόνο ε, σύστημα καταχώρησης εισόδου και σε εποχές κρίσης που στην Ελλάδα και στην Ισπανία και αλλού ε, επιβάλλουμε συνέχεια προγράμματα αλητότητας, όπου κόβουμε συντάξεις, όπου ο κόσμος ε, δεν έχει πρόσβαση σε ένα καλό σύστημα γιατρικής περίθαψης, ε, πώς μπορούμε να πούμε στις χώρες αυτές, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιρλανδία, ότι θα δώσουμε ένα δισεκατομμύριο ευρώ για ένα σύστημα συλλογής στατιστικών. Πώς θα το πούμε αυτό σε όλους ε, τους ε, νέους άνεργους. Ε, πάνω από το 50% των νέων σε κάποιες περιοχές είναι άνεργοι, αλλά εμείς προτιμούμε να δώσουμε ένα σωρό χρήματα για ένα τέτοιο σύστημα, τη στιγμή που δεν γνωρίζουμε καλά-καλά τη χρησιμότητα του συστήματος αυτού. Δεν ξέρουμε καλά-καλά εμείς τι θέλουμε από το σύστημα αυτό. Η κυρία Σόμερ, όπως και τα κράτη-μέλη, Η κυρία Σόμερ ζητεί το σύστημα αυτό να χρησιμοποιηθεί και για την καταπολέμηση του εγκλήματος ε, ήδη από την αρχή. Ε, αυτό βέβαια απαιτεί τα δαχτυλικά αποτυπώματα των ταξιδιωτών ε, αυτή τη στιγμή. Έχουμε όμως παρόμοια τέτοια συστήματα στην Γερμανία κατά την εισαγωγή του ηλεκτρονικού διαβατηρίου ηθελημένα ε, ε, ε, παρετηθήκαμε από την ιδέα μιας βάσης δεδομένων διότι δεν θεωρήσαμε ότι θα είναι χρήσιμο και στην Γαλλία ε, θεωρήθηκε αντισυνταγματική η ύπαρξη ε, βάσει δεδομένων με δαχτυλικά αποτυπώματα όλων των πολιτών ε, και για λόγους προστασίας δεδομένων και οι κάτω χώρες δεν δημιούργησαν ένα τέτοιο σύστημα και εμείς τώρα θέλουμε να δημιουργήσουμε μια τέτοια βάση δεδομένων για υπηκόους τρίτων χωρών και για αυτούς τους ανθρώπους ισχύουν τα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων. Γιατί λοιπόν θέλουμε να κάνουμε διακρίσεις και να Επιβάλλουμε σε αυτούς ε, συλλογή δεδομένων ε, που απαγορεύεται να γίνεται για Ευρωπαίους πολίτες. Και ε, θεωρούμε ότι εκ των προτέρων ότι είναι πιο εγκληματίες από εμάς και Κομισιόν τόνισε ότι η συλλογή ε, ε, ε, δαχτυλικών αποτυπωμάτων αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να γίνει και ότι θα οδηγήσει σε σημαντικές καθυστερήσεις. Δεν καταλαβαίνουμε λοιπόν πώς μπορούμε να συμπεριλάβουμε από την αρχή τα βιομετρικά στοιχεία. Δεν έχουμε εμπειρίες από το σύστημα πληροφόρησης για τις θεωρήσεις. Από το πιλωτικό πρόγραμμα 2 ξέρουμε ότι ότι ε, χρειάζονται δύο λεπτά περίπου για τα... τρία λεπτά απαιτούνται για τα δακτυλικά αποτυπώματα. Ε, αυτό σημαίνει τρία λεπτά παραπάνω στις, ε, στα σύνορα, σημαίνει δηλαδή μεγάλες ουρές και αν έχουμε περισσότερους ταξιδιώτες στο μέλλον, τη στιγμή που τώρα ήδη οι διευθύνσεις των αεροδρομίων λένε ότι δεν έχουν αρκετά χώρο για τους ανθρώπους που περιμένουν, στο μέλλον τι θα κάνουμε με αυτούς οι τουρίστες, οι σπουδαστές, ε, οι επιχειρηματίες. Ε, θέλουμε ε, όλους αυτούς να τους αφήσουμε να περιμένουν σε μεγάλες ουρές. Τι θα γίνει με τον χώρο γνώσης και καινοτομίας στην Ευρώπη. Η Κομισιόν λοιπόν στην μελέτη επιπτώσεων δεν αναφέρεται στο θέμα αυτό. δεν ασχολείται ούτε με τα δαχτυλικά αποτυπώματα, ούτε με τα θεμελιώδη δικαιώματα, ούτε με τις ε, καθυστερήσεις ε, και το χρόνο αναμονής ε, που θα υπάρξει. Αν θέλουμε να αυτοματοποιήσουμε από την αρχή το σύστημα, θα πρέπει να εξετάσουμε και τις συνέπειες για την πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου. Ε, αυτό δεν αναφέρεται καθόλου στη μελέτη επιπτώσεων και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να γίνει πολύ προσεκτική ε, αξιολόγηση. Τι συνέπειες έχει αυτό για την προστασία των δεδομένων, ε, για τον χρόνο αναμονής για την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων. Εάν λοιπόν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια πολιτική, θα πρέπει να εξετάσουμε τις συνέπειες και χρειαζόμαστε τουλάχιστον μια κοινοβουλευτική μελέτη επιπτώσεων που είναι επιθυμία και ε, ε, που θα εξετάσει τις επιθυμίες και της εισηγήτριας και των κρατών μελών. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι συνέπειες για τα αεροδρόμια, για τα θεμελιώδη δικαιώματα, για την ευρωπαϊκή οικονομία. Ελπίζω να μπορεί να γίνει αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Απλώς θα επικεντρωθώ στο σύστημα εισόδου-εξόδου, το οποίο προφανώς όπως και άλλοι συνάδελφοι καλωσορίζω. Καλωσορίζω την εισαγωγή ενός τέτοιου συστήματος, διότι προφανώς βοηθά να μειώσουμε, να καταπολεμήσουμε την λάθρο Επίσης, επιτρέπει στα κράτη-μέλη να λάβουν καλύτερη μέρημνα για την αντιμετώπιση ενός τέτοιου φαινομένου. Ωστόσο υπάρχουν κάποια μικροπροβληματάκια. Όχι για το ζήτημα αυτό καθεαυτό, αλλά για την πρακτική διοργάνωσή του. Έχω άμεση εμπειρία του, των συστημάτων IT και του πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αξιοποιηθούν και σε πολιτικό επίπεδο και εκτός. Τη δεκαετία του 90 ήμουν ένας από τους πρώτους που χρησιμοποίησα στη νομική μου εταιρεία για τα λογιστικά το σύστημα Word και την ε, επεξεργασία των ε, δεδομένων κατά αυτόν τον τρόπο. Ε, η αποθήκευση 100 MB, στοιχείων 100 MB, έπρεπε να γίνει σε μια αίθουσα 8 φορές μεγαλύτερη από την αίθουσα στην οποία βρισκόμαστε, με τεράστια κλιματιστικά μηχανήματα για να υπάρχει συνεχώ ο κατάλληλος αερισμός. Λοιπόν, όπως είδαμε εδώ, ε, γύρονται, ε, γύρονται ζητήματα τα οποία έχουν σχέση και με παρόμοιες προσπάθειες που έγιναν και στο Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού. Τέτοια συστήματα προσπάθησαμε να καταρτήσουμε για το σύστημα υγείας, για τα συνταξιδικά ταμεία και βεβαίως ναι και για την ενέργεια των συνόρων. Το κόστος όλων αυτών των προσπαθειών μπορεί πραγματικά να φύγει και να ξεφύγει εκτός του ελέγχου μας. Εν ώψη λοιπόν των ε, σημαντικών επενδύσεων που θα απαιτηθούν για να μπορέσει να γίνει πράξη και να λάβει σάρκα και τα ένα τέτοιο σύστημα εισόδου και εξόδου αλλά και αυτό τη καταχώρηση ταξιδιωτών θα ήθελα να καταλάβω από το Ταμείο για την Εσωτερική ε, Ασφάλεια από το 2014 στο 2020 διαθέτουμε κονδύλια, μπορούμε να ελέγξουμε το κόστος ή θα σφάλουμε τελείως τον αρχικό υπολογισμό του κόστους. Θα μπορέσουμε να ελέγχουμε την εξέλιξη των συμβάσεων ε, στις οποίες ε, θα, με τις οποίες θα συμβληθούμε ως προς τα βιομετρικά δεδομένα και την πρόσβαση σε αυτά των ε, διοκτικών αρχών θα έπρεπε να είναι προφανώς μέρος του συστήματος εισόδου και εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευθύς εξ αρχής και όχι να χρειαστεί ε, να επεκταθούν οι σκοποί και το πεδίο των αρχικών σκοπών αργότερα. Δεν είναι ωραίο να προσθέτουμε πράγματα ε, στη συνέχεια. Να δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το Eurodac, όπου εκεί έχουμε αντιμετωπίσει παρόμοιες δυσκολίες. Αλλά η ανάγκη για τη χρήση των βιομετρικών δεδομένων νομίζω είναι προφανής και θα πρέπει να λάβουμε την ε, ανάλογη απόφαση. Αυτό που αρκεί να κάνουμε είναι να δούμε τι διδάγματα έχουμε από την εμπειρία άλλων, ιδίω των ΗΠΑ. Εκείνοι τα βιομετρικά δεδομένα τα εισήγαγαν με τεράστιο, απίστευτο κόστος. Βέβαια είναι πολύ μεγαλύτερο το εγχείρημα των ΗΠΑ, αλλά μιλάμε για δισεκατομμύρια δολάρια και νομίζω ότι δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να δουν τι πραγματικά ωφέλη μπόρεσαν να αντλήσουν από αυτό το σύστημα. Δεν θέλω λοιπόν να ακουστώ απλώς σκεπτικιστής και διστακτικός. Δεν είμαι πραγματικά σκεπτικιστής, σας το ορκίζομαι, αλλά πρέπει να ακουστούν αυτές οι αμφιβολίες και αυτοί οι ενδιασμοί. Επί της αρχής, θεωρητικά, συμφωνώ απολύτως, 100%. Ε, θα ήταν υπέροχο αν γινόταν πράξη όλο αυτό. Όμως πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ καλά τους περιορισμούς που έχουμε από την πλευρά του προπολογισμού και να λάβουμε υπόψη τις εμπειρίες άλλων. Πρέπει να μπορούμε να προβλέψουμε τι αποτελέσματα θα προκύψουν. Συγγνώμη που είμαι λίγο αρνητικός πρόεδρε, αλλά πρέπει να είμαστε πραγματικά ιδιαίτερα προσεκτικοί με τέτοια θέματα. Ευχαριστούμε πρόεδρε. Κύριε Κίρκοπ. και άλλοι συνάδελφοι θέλουν να παρέμβουν. Η κυρία Ματιού. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα έλεγα να προσπαθήσετε από εδώ και μπρος να είστε σύντομοι όλοι οι υπόλοιποι, διότι πραγματικά έχουμε καθυστερήσει. Έχουμε και άλλο σημείο πριν την συνάντηση των συντονιστών. Νομίζω, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, η αυτή μέτρων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά θα πρέπει να βελτιωθεί σε κάποια σημεία τη Ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά το κόστος, όπως είπε και ο κύριος Ένθιου, 300 εκατομμύρια ευρώ νομίζω να φέρετε, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, νομίζω όντω θα πρέπει να περιοριστεί το κόστο αυτού του εγχειρήματο. Είναι όμω απαραίτητο. Τα εφή σύνορα χρειάζονται. Όλοι οι πολίτε παραπονούνται για τα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί οι ίδιοι ε, παραπονιόμαστε για τι ελλείψει και τα κενά παρουσιάζονται στον έλεγχο των σύνορων μα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να αναλάβουμε εδώ κάποια μέρημνα. Ε, θα πρέπει να το εξετάσουμε το θέμα αυτό. Βεβαίω, στο επίπεδο του συστήματος καταχώρησης ταξιδιωτών. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ίσως να μην είναι η καταλληλότερη γιατί θα μπορούσε να προτείνει κάτι περισσότερο στην κατεύθυνση των όσων κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Θα ήταν πιο συνετό πιστεύω και η δική τους προσπάθεια δίνει καλά αποτελέσματα νομίζω. Γιατί να μην βασιστούμε σε αυτό. Το κόστος ε, κατά πάσα πιθανότητα θα ήταν πιο περιορισμένο και όσοι έχουν κάνει οι Αμερικανοί είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα. Όσο για τον κανονισμό που αφορά το σύστημα εισόδου και εξόδου, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε το κατά πόσον αυτό το ντοσχέ θα εμπλέξει και τις αστυνομικές δυνάμεις θα πρέπει να έχουν πρόσβαση ευθύς εξ αρχής στα βιομετρικά δεδομένα εκείνη. Αλλά εδώ να μην ξεχνάμε και για το σεβασμό της χάρτας των θεμελιωδών δικαιωμάτων ας μπορούν να έχουν πρόσβαση από την αρχή μεν, αλλά δεν ε, έχει κανένα νόημα να θεσπίσουμε ένα τέτοιο σύστημα αν δεν μπορούν από την αρχή να έχουν πρόσβαση οι αστυνομικές δυνάμεις. Και χάρη σε αυτό το πακέτο των, των συνόρων δεν μπορούν να καταπολεμήσουν την ε, λαθρομετανάστευση. Μου φαίνεται πραγματικά άκρο σημαντικό αυτό ε, από την αρχή της συζήτησή μας. Διότι πραγματικά όλα αυτά μπορούν να εξυπηρετήσουν, να διευκολύνουν την ε, αναχέτηση της ε, λαθρομετανάστευσης. Όσο προς τις ε, ουρές αναμονής και όλα τα σχετικά προβλήματα, αυτά θα τα δούμε. Το θέμα είναι να υπάρχει ρευστότητα. Ρευστότητα η οποία θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί ως θέμα από το πρώτο πακέτο. Οι ταξιδιώτες που έρχονται συστηματικά από τρίτες χώρες χάρη στον πρώτο κανονισμό θα ταξιδεύουν ε, πιο άνετα. Δεν ανησυχώ λοιπόν ιδιαίτερος ως προς το πρόβλημα που έθεσε η κυρία Κέλλερ. Ρομέρο. Κυρία Ρομέρο. Πρόεδρε, Νομίζω ότι η κυρία Πλερ ζήτησε πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Για το σύστημα, για το πρόγραμμα καταχώρησης ταξιδιωτών ε, πιστεύω ότι ζητείται από τους ανθρώπους ε, να δώσουν πάρα πολλά στοιχεία για τον εαυτό τους ε, και ε, θα πρέπει να εξετάσουμε μήπως γίνεται διάκριση εις βάρος κάποιων με αυτήν την διευκόλυνση της πρόσβασης. Η ομάδα του άρθρου 29 ανέφερε ότι δεν θα ελέγχουμε όλους τους ταξιδιώτες. Ελπίζω όμως αυτό να μην οδηγήσει ε, στο στο να μην ε, υπάρχει αυτό μόνο για τα ε, αεροδρόμια και τελικά να έχουμε ελέγχους παντού αλλού. Επίσης, όσον αφορά τις σφραγίδες, ήδη απαντήσατε ε, στο πρόβλημα αυτό τη στιγμή που έχουμε όλο και περισσότερες ε, ε, συμφωνίες διευκόλυνσης θεωρήσεων. Έτσι λοιπόν δεν θα έχουμε όλα τα προβλήματα που αναφέρονται εδώ πέρα. Το θέμα της λαθρομετανάστευσης, το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν έχουμε δεδομένα, αυτοί που παραμένουν περισσότερο από, από όσο πρέπει είναι όλοι οι εγκληματίες και τρομοκράτες. Δεν έχουμε τέτοια δεδομένα, ωστόσο γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που παραμένουν παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επειδή βρίσκονται εδώ παράνομα, ε, τους εκμεταλλεύονται στην αγορά εργασίας ε, ε, και αλλού. Εποφελούνται δηλαδή άλλοι από αυτές τις παράνομες παραμονές. Και εάν γνωρίζω ότι κάποιος ε, έχει παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα τι κάνω τις πληροφορίες αυτές ε, Θα γνωρίζω πού βρίσκεται. Η κυρία Σόμερ είπε ότι δεν χρειαζόμαστε μόνο τα φιλικά αποτυπώματα, χρειαζόμαστε και φωτογραφία. Ε, χαίρομαι που έτσι θα μπορούμε να έχουμε και βίντεο παρακολούθηση παντού. Αυτό θέλουμε. προφανώς όχι. Ε, λέμε ότι το σύστημα αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε και για άλλους ε, στόχους ε, και αναρωτιέμαι εγώ μήπως ο μεγάλος αδερφός ήδη βρίσκεται εδώ μεταξύ μας. Και βρίσκω γελία τη συζήτηση που έχουμε αυτή τη στιγμή διότι Ξέρουμε, πώς, ε, ξέρουμε τι κάνουν τα κράτη που ενδιαφέρονται να συλλέξουν συγκεκριμένε πληροφορίε, και όσον αφορά το κόστο, που είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο ε, γνωρίζουμε από τι εμπειρίε μα ότι ώρα θα είναι πιο ακριβά από αυτό. Ε, βρίσκω ότι είναι όλα αυτά τελείως δυσανάλογα τη της κατάστασης σε κάποια κράτη-μέλη, δεδομένων των κοινωνικών προκλήσεων και δεδομένης τη χρήση του προγράμματο. αυτού. Βρίσκω ότι είναι τελείω δυσανάλογο το κόστο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, να ευχαριστήσω την Ρενάτε Σόμερ και τον κύριο Έντσου για τα έγγραφα εργασίας που έχουν ετοιμάσει και πραγματικά συμμερίζομαι τις απορίες τους. Τα χρειαζόμαστε τα συστήματα αυτά. Τι προστιθέμενη αξία θα μας προσφέρουν. Τα συστήματα αυτά είναι ο καλύτερος τρόπος για να, ασχολ... για να ξέρουμε τις λύσεις που μας λείπουν. Κατανοώ ότι το κείμενο του κυρίου, της κυρίας Σόμερ είναι πιο αισιόδοξο και πιο διστακτικό εκείνο του κυρίου Ένσου. Εγώ θα έλεγα ότι καλύτερα θα ήταν να είμαστε περισσότερο συνετοί ως προς τα συστήματα αυτά. Περισσότερο επιφυλακτικοί. Και έχω να θέσω πέντε ερωτήσεις. Πέντε ζητήματα. Πρώτον, τι θα μας προσφέρουν αυτά τα συστήματα. Όπως ήδη είπαν κάποιοι συνάδελφοι, και ως προς τις αρχές προστασίας δεδομένων, τι μας προσφέρουν πληροφορίες που αφορούν τους παρανόμους διαμένοντες. Όμως δεν έχουμε κανενός είδους πληροφορία για τον γεωγραφικό τους εντοπισμό. Δεν έχουμε καμία νέα λύση για να διευκολύνουμε τις διαδικασίες επιστροφής. Δεν έχουμε καμία νέα λύση στην περίπτωση όπου ένα τρίτο κράτος δεν ε, φαίνεται συνεργάσιμο για την επιστροφή των ε, ανθρώπων αυτών. Άρα η αίσθησή μου είναι ότι αυτό που θα μας προσφέρει αυτό το νέο σύστημα δεν είναι και κάτι τόσο φοβερό. Το δεύτερο ζήτημα, κάτι που έθεσε ήδη ο κύριος Κίλκοπ. Θα λειτουργήσει όλο αυτό. Διότι όπως είδαμε οι Ηνωμένε Πολιτείε της Αμερικής εδώ και μία δεκαετία έχουν δαπανίσει αμύθιτα ποσά και ούτε εκεί λειτουργεί το σύστημα. Εδώ γιατί θα λειτουργήσει. Γιατί. Περιμένουμε και φανταζόμαστε ότι θα πετύχει σε εμά. Τρίτο ερώτημα. Τι κόστος θα υπάρξει. Άκουσα τον κύριο Έντσου. Και σίγουρα το 1,1 μπορεί να φτάσει το 1,3 εύκολα. Όμω θυμάμαι την πρώτη φορά που πρότεινε το ΣΥΣ2 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συζητούσαν για 23 εκατομμύρια. 23 εκατομμύρια. Τελικώ το κόστο έφτασε τα 165 εκατομμύρια. 165. Εάν θέλουμε να προσθέσουμε τα χρήματα μάλιστα που χρειάστηκε να δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις φορήσει διαχείριση των εξωτερικών σύνορων για να τους βοηθήσει, μιλάμε για 95 εκατομμύρια ήδη. Συνολικά μιλάμε για κόστος 250 εκατομμύρια για το ΣΕΣ2. Ενώ ξεκινήσαμε από ελάχιστα. Εδώ για πόσα δις μιλάμε πέντε φορές περισσότερα από ό,τι από το ΣΥΣ 2. Και είναι μόνο η πρώτη φάση. Ποιο θα είναι το τελικό κόστος. Πέντε δις. Δεν νομίζω να απαντήσει κανείς αυτό. Τέταρτη ερώτηση. Ξέρουμε τι μπορούμε ήδη να κάνουμε Και το ανέφερε αυτό και η ομάδα εργασία του άρθρου 29. Τώρα μόλις περάσαμε στη δεύτερη γενιά του ΣΕΣ 2. Και τώρα υλοποιείται και παίρνει σάρκα και οστά το σύστημα ΒΙΣ. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε για να αποτιμήσουμε τι ωφέλη αντλούμε από αυτά τα συστήματα. Θέλουμε να αποφύγουμε τις επαναλήψεις και τις επικαλύψεις. Δεν το βρίσκω συνετό να δαπανίσουμε τέτοια ποσά για να δημιουργούμε νέα συστήματα, ενώ κατά πάσα πιθανότητα τα συστήματα που ήδη έχουμε μπορούν να μας καλύψουν. Τελευταία παρατήρηση. Προστασία δεδομένων. Δεν θα επαναλάβω όσα είπαν οι συνάδελφοι. Τα είπαν και αρχέ προστασία των δεδομένων. Πραγματικά εδώ υπάρχουν σοβαρέ ε, ανησυχίε για το πώ θα προστατεύονται τα δεδομένα ω προ τα συστήματα αυτά. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω, Πρόεδρε, με μία σημείωση. Ήδη από το Φεβρουάριο του 2012, σε μια διάσκεψη που οργάνωσε, οργάνωσε η τότε Προεδρεύουσα Δανική ε, Προεδρεύου του Συμβουλίου στην Κομεχάγη για την καινοτομία στον έλεγχο των συνόρων, Πήγαμε τον κύριο Ένσιο και την, και την κυρία Κέλλερ και ακούστηκαν σοβαροί ενδιασμοί για το πακέτο αυτό των εφιών συνόρων τότε είχα αναφέρει ότι υπάρχουν άλλες προτεραιότητες, άλλες προτεραιότητες που η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει γρήγορα. Επέμεινα στην αναβολή εξέτασης του συστήματος ε, του, του πακέτου ευθείων συνόρων. Ε, είπα ότι ήδη υπάρχουν μέτρα και τεχνολογικές πρακτικές λύσεις που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε ένα μεγάλο και ευρύτερο σκηνικό αξιοποίησης των ε, τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εμείς περάσαμε όλη την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο μιλώντας ε, για τον έλεγχο της μετανάστευσης, ε, το SIS, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας κτλ. κτλ και τα τμήματα του προϋπολογισμού που ανήκουν σε, αυτές τις, ε, ε, σε αυτά τα θέματα έχουν απορροφηθεί ήδη για θέματα SIS ε, και για τα συστήματα κοινής χορήγησης ασύλου κτλ. Υπάρχουν άνθρωποι βέβαια οι οποίοι έρχονται στην Ευρώπη για πάρα πολλούς λόγους και είναι σαφές ότι θα πρέπει να ελεγχθούν, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να δούμε τι αιτίες βρίσκονται πίσω από την ε, περαιτέρω παραμονή αυτών των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως εκεί μπορούμε ακριβώς να σκεφτούμε κάποια πράγματα αρκετά ευφυή για να βρούμε μία ε, λύση. Εμείς αυτή τη στιγμή αλλάζουμε ένα σύστημα κατασταλτικό θα έλεγα με ένα άλλο σύστημα το οποίο είναι φιές υποτίθεται, ηλεκτρονικό το οποίο όμως ε, νομίζω ότι δεν θα λύσει τα προβλήματα. Εμείς ταυτίζουμε ουσιαστικά αυτόν ο οποίος παραμένει πέραν της αρχικής περίοδου ε, πολίτη από τρίτη χώρα με τρομοκράτη, τον παράνομο μετανάστη τον ταυτίζουμε με κακοποιό. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε μία πρωτοβουλία και να προσπαθήσουμε να δούμε τι λόγοι βρίσκονται πίσω από αυτόν τον παραμένοντα και να δούμε τι διαφορές υπάρχουν ανάμεσα στους πολίτες των χωρών μας και τους πολίτες των χωρών αυτών όταν έρχονται ε, στις ε, πατρίδες μας, να δούμε τι έφυσαν πίσω τους, τις συνθήκες εργασίας, τις κοινωνικές συνθήκες, τις συνθήκες υγείας και υγιεινής. Δεν μπορούμε να εφαρμόζουμε συνεχώς προγράμματα και συστήματα καταστολής, προγράμματα και συστήματα τα οποία θεωρούν ότι οι ξένοι οι μετανάστες είναι είτε τρομοκράτες είτε κακοποιοί. Νομίζω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάψει να παρουσιάζει τέτοιου είδους σχέδια συστηματικά. Η κυρία Κοράτσα. η πρόταση της Επιτροπής και οι προτάσεις των δύο εισηγητών έχουν ενδιαφέρον. Βέβαια υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία παραμένουν χαίνοντα στην παρούσα φάση. Έχει μεγάλη σημασία να προσπαθήσουμε να ε, δώσουμε την ασφάλεια που θέλουν ε, οι πολίτες μας και να υπάρχει ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου στα σύνορα. Ήδη έχουμε ένα τέτοιο σύστημα, η νέα γενιά και του SIS και τα λοιπά. Και θα συμφωνήσω με τον κύριο Κοέλιο ότι καλό θα ήταν να προσπαθήσουμε να δούμε πρώτα πώς δουλεύει το σύστημα αυτό το πληροφορικό καταρχάς και ε, αν μπορούμε να το βελτιώσουμε και να το αναπτύξουμε. Ένα δεύτερο θέμα είναι το θέμα του κόστους και της αποτελεσματικότητας της χρήσης συγκεκριμένων πιστώσεων και σε επίπεδο δημοσιονομικό και σε επίπεδο γραφειοκρατικού άχθους για τα κράτη-μέλη, τα μικρά ιδιαίτερα, τα οποία έχουν εκατοντάδες σημεία εισόδου και να μην αναφερθώ στα θέματα τα προξενικά, στα προξενία, που ε, θα πρέπει να έχουν τεράστιες υποδομές για να μπορούν να χειριστούν τα συστήματα καταγραφής αιτήσεων. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν να δούμε ακριβώς και τα θέματα τα οποία έθεσαν ε, οι εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Επιθεωρητών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να μελετήσουμε περισσότερο τις δυνατότητες που υπάρχουν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και να δούμε ακριβώς τι ωφέλη θα έχουμε σε επίπεδο ασφάλειας. Έχει σημασία επίσης να θεωρήσουμε ότι το σύστημα αυτό θα πρέπει να είναι πλήρως εθελοντικό. Κάποιες χώρες ε, μπορεί να το επιθυμούν και να θέλουν να το χρησιμοποιήσουν, κάποιες άλλες να θεωρούν ότι δεν θα έχουν ε, το απαιτούμενη τη σωστή σχέση ε, κόστους ωφέλους και θέλουν να είναι το σύστημα αυτό στην εφαρμογή του πιο ευέλικτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι ο συνδυασμός δημοσίων αρχών και τεράστιων προγραμμάτων πληροφορικής είναι ένας ευτυχής συνδυασμός. Δεν γνωρίζω πολλά παραδείγματα τεράστιων προγραμμάτων που έχουν πετύχει πάντα μένουν από χρήματα, πάντα δεν φτάνουν να καλύψουν τις προσδοκίες, αλλά από ό,τι φαίνεται όμως αυτό δεν μας γίνεται μάθημα και κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει προτάσεις σαν και αυτές που, γίνουν, που κάνουν στην τηλεόραση, προσπαθούν να σας πουλήσουν νέα μηχανήματα τα οποία θα λύσουν τα προβλήματα που δεν ξέρατε ότι είχατε. Νομίζω ότι σε εποχές οικονομικής ιδιαίτερα κρίσης υπάρχουν καλύτεροι τρόποι για να ξοδέψουμε ακριβώς αυτό το 1 δις 100 εκατομμύρια που στο τέλος θα γίνει 5. Αν δείτε το τι γίνεται στη Νότια Ευρώπη με 60% ανεργία των νέων η απάντηση που θα δώσουμε είναι αυτό που λέει η Επιτροπή. Και όπως είπε πολύ σωστά ο Κοέλιο, η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή και στις Ηνωμένε Πολιτείες. Ήδη και στις Ηνωμένε Πολιτείες δεν δουλεύει το σύστημά τους. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι εμείς θα το κάνουμε αυτό. Πώς πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πιο αποτελεσματική από την Αμερικανική Υπηρεσία, Υπουργική Υπηρεσία Ασφαλείας ε, της ε, χώρας. Και θα έλεγα στον κύριο Κύρκο που όποιος έφυγε όμως ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Η εταιρεία σαν παράδειγμα που είχε δημιουργήσει το σύστημα απελήθη κόστισε πάρα πολλά στο δημόσιο. Ήταν μια τεράστια σε επίπεδο ε, εξοπλισμού προσπάθεια και απαιτείται περισσότερη προσοχή. Και θα ήθελα πρώτα λοιπόν να μου δώσουν την εξής απάντηση στο εξής ερώτημα. Ποια είναι τα προβλήματα που θέλετε να λύσετε. Αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι θα διευκολύνουμε λέει τα ταξίδι για τους Ευρωπαίους και θα μικρύνουν οι ουρές στα αεροδρόμια. Τα έχουμε ακούσει αυτά ξανά και στην περίπτωση του PNR ή το Trusted Traveler, ο έμπιστος ταξιδιώτης. Δεν ξέρω αν είδατε να μικραίνουν οι ουρές στα αεροδρόμια πουθενά. Λοιπόν και για ε, να μπορούμε να βρούμε ακριβώς αυτούς οι οποίοι παραμένουν μετά από τη λήξη. Α, κοιτάξτε, αυτό δεν γίνεται όταν μπαίνουν στα σύνορα. Έτσι και αλλιώς περνώντας τις χώρες μας μπορεί να πάνε παντού. Και στο τέλος λένε ότι ίσως κάποια στιγμή κάποτε η δικαστική υπηρεσία, η αστυνομική υπηρεσία και οι ε, υπηρεσίες ασφαλείας γενικότερα θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα. Όχι, αυτό δεν πρέπει να γίνει. Δεν έχω ακούσει καμία ουσιαστική δικαιολογία για τη συγκεκριμένη πρόταση και η πρόταση αυτή πρέπει να διαγραφεί. Λοιπόν, αυτά. Ε, επανέρχομαι στους... Α, όχι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ορίζουμε την ευκαιρία αυτή. Παρακαλώ σύντομα τις παρατηρήσεις σας, γιατί έχουμε καθυστερήσει, έχουμε κι άλλη συζήτηση, κι άλλο θέμα να εξετάσουμε. Ναι, ναι, θα είμαι πολύ σύντομος, γιατί έρθηκαν πάρα πολλά ερωτήματα και ζητήματα και καλώς ορίζουμε το λίγο χρόνο που μας δίνεται για να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε. Κατά πρώτον, νομίζω, ένα από τα συνολικά ζητήματα είναι το κατά πόσον χρειαζόμαστε αυτά τα συστήματα και αν τα συστήματα αυτά είναι αναλογικά. Η απάντησή μας είναι προφανώς καταφατική. Ναι, αλλά όχι γιατί απλώς ε, χρειαζόμαστε ένα ακόμη ακριβό σύστημα σε συνθήκε χρηματοπιστωτικής και οικονομική κρίση. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά πώς έχει το οικονομικό ε, τοπίο και είμαστε πολύ ταπεινοί για τι ε, προηγούμενε προσπαθίες μας για να αναπτύξουμε συστήματα IT όπω το SIS2 και το VIS. Ε, Όντω ε, έχουμε αντλήσει κάποια διδάγματα από την εμπειρία των συστημάτων αυτών που μας δείχνουν πώς, καλύτερα να, πώς να ετοιμαζόμαστε καλύτερα για τέτοιου είδους προτάσεις και για να αντιμετωπίσουμε την αύξηση του κόστους. Η πείρα μας μας έχει διδάξει. Και ακριβώς αυτό μας οδήγησε και ως προς το κόστος και το περιεχόμενο στο να υποβάλουμε ακριβώς αυτή την δέσμη μέτρων για τεφή σύνορα. Ποιος είναι τώρα Ποιο είναι το πεδίο, ποιο είναι ο βασικό σκοπό. Οι περισσότερε απόψει και παρατηρήσει εντοπίστηκαν στη λαθρομετανάστευση και την αναχέτησή τη. Κατά πόσο τα συστήματα αυτά μπορούν να μα το επιτρέψουν αυτό. Ένα ζήτημα που παραβλέπετε ότι ο πρωταρχικό σκοπό ενό τέτοιου συστήματο, του συστήματο καταχώρηση ε, των ταξιδιωτών λόγου χάρη, είναι να διευκολύνουμε του συνοφύλακε. Αφήστε τώρα όλε τι άλλε εικασίε και υποθέσει. Όπω είπε ο κ. πρέπει να δούμε αν είναι ορθό ή όχι κάτι ή αν πιστεύουμε όχι τις εικασίες όμως βάσει των σημερινών αριθμητικών στοιχείων, οι συνοριοφύλακέ μας έχουν μεγάλες δυσχέρειες προκειμένου να υλοποιήσουν τα όσα επιβάλλει το κεκτημένο του Σέγγεν. Και εδώ έχω και ακόμη μερικέ παρατηρήσει ε, που έκαναν κάποιες από, κάποια από τα μέλη της Επιτροπής για τα εξωτερικά σύνορα και το αν οι συνοριοφύλακε ε, καταγράφουν σωστά τι ε, εισόδους και εξόδους Ναι, είναι ένα ζήτημα αυτό. Σήμερα, κάθε μέρα σε κάθε σημείο ελέγχου των συνόρων, θαλάσσιο, χερσαίο ή αεροπορικό, καταγράφουν τα πάντα σε χαρτί όμως, με σφραγίδες και στυλό. Αυτό χρειάζεται χρόνο. Χάνει χρόνο και ο συντοφύλακα και οι ταξιδιώτε και είναι πολύ παροχημένος τρόπο να αντιμετωπίζουμε ένα τέτοιο θέμα που θέλουμε να λάβει μια καλύτερη αντιμετώπιση, δηλαδή τη διαχείριση των συνόρων μας. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο να κατηγορήσουμε, να κυνηγήσουμε, να καταδιώξουμε τους παρανόμως στην Ευρώπη, ούτε θέλουμε να τους βάλουμε κανένα, ε, καμιά στάμπα στο κούτελο. Όχι, θέλουμε απλώς να διαχειριστούμε καλύτερα τα σύνορά μας. Κάτι ε, στο οποίο ούτως ή άλλως Βάσει των σημερινών μας στοιχείων βλέπουμε ότι δύσκολα το διαχειρίζονται οι σύνοριοφύλακες οι ίδιοι. Είναι σοβαρότατο σκοπό αυτό. Σίγουρα υπάρχουν ενδιασμοί, αλλά είναι σημαντικό το να ξέρουμε ποιο είναι παρανόμο διαμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην περιοχή, στον χώρο του Σέγγεν, είναι σημαντική, ε, σημαντικό στόχο. Θα πρέπει οι αρχέ να δουν πώ θα υλοποιήσουν μετά την ε, πολιτική μετα... την ε, πολιτικη αναχετηση τη λαθρομετανάστευση που ήδη υπάρχει. Η πολιτική αυτή προβλέπεται. Δεν είναι κάτι που θα το προβλέψουμε τώρα. Οι παρανόμω διαμένοντε είναι λαθρομετανάστες από τη στιγμή που γίνονται παρανόμως διαμένοντες ε, εξισούνται με τους μετανάστες. Τώρα, άλλο είναι αν θα το δούμε στο ευρωπαϊκό ή στο εθνικό επίπεδο πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Αλλά θα ξέρουμε πού να τους βρούμε. Εκτός από την καλή διαχείριση λοιπόν των σύνορων, το σύστημα αυτό θα δίνει στις αρμόδιες αρχές ένα σημείο αφετηρίας για να μπορέσουν να αναπτύξουν τις πολιτικές που χρειάζονται, για να αντιμετωπίσουν τη λαθομετανάστευση βάσει των όσων ήδη διαθετούν ως εργαλεία. Άκουσα αρκετές παρατηρήσεις και από την Αρχή Προστασία των Δεδομένων και από την Ομάδα Εργασία του Αρχικού 29 και κάποιου από του συναδέλφου σα εδώ για τη δημιουργία μια τεράστια βάση δεδομένων. Με δεδομένα για όλου του πολίτε και αν αυτό είναι αναλογικό. Και γιατί να το κάνουμε κάτι τέτοιο. Αλλά να σα επιστήσω εδώ την προσοχή σα στο εξή. Περίοδο στήριξη των δεδομένων. Στο κείμενο έχουμε προτείνει, νομίζω, κάτι πολύ λογικό και αναλογικό, ώστε να ε, καλύψουμε ε, και την ε, συλλογή διοντρικών δεδομένων και την πραγματική καταγραφή των δεδομένων. Είναι σύντομη η περίοδος αυτή, είναι σύντομη η διάρκεια και από τις αρχές και από τους ε, συνοφύλακες. Τη στιγμή που εκπνέει η διάρκεια αυτή, τα δεδομένα διαγράφονται από το σύστημα. Η περίοδος λοιπόν τήρησης των δεδομένων, όπως την έχουμε προβλέψει στην πρότασή μας, είναι αυτή η αυτή εγγύηση για το ότι τα δεδομένα δεν θα τηρηθούν περισσότερο χρόνο, δεν θα αποθηκεύονται περισσότερο από ότι είναι απολύτω απαραίτητο για τι ανάγκε του συστήματο. Για του παρανόμου διαμένοντε η περίοδο αυτή θα μπορούσε να παραταθεί, αλλά για λόγου που έχω ήδη εξηγήσει. Μέχρι να δουν τι σύστημα θα εφαρμόσουν οι αρμόδιε αρχέ. Το κόστο τώρα. Πολλέ ερωτήσει τέθηκαν και σωστά νομίζω, πολλέ ερωτήσει τέθηκαν για το κόστο. Κατά πρώτον, εμπιστευόμαστε τα αριθμητικά στοιχεία τη πρόταση. Καταρχά, και πραγματικά σωστά το λέτε κι εσεί, πραγματικά έχουμε κάνει πάρα πολλές συγκριτικές μελέτες για το κόστος και σε σχέση με το ΣΕΣ2 και το ΒΙΣ. Και πάλι θα έλεγα ότι η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική. Και είναι διαφορετική ακριβώς λόγω της πείρας που έχουμε αντιλήσει από το ΣΥΣΔΙΟ. 2 Ναι, το ΣΥΣ αρχικά είχε προβλεφθεί για, τα, για 53 εκατομμύρια και έφτασε 400 δις. Λοιπόν, Γι' αυτό τώρα έχουμε προβλέψει 500 εκατομμύρια. Διότι αυτή τη φορά δεν βασιζόμαστε στις ίδιες υποθέσεις και προβλέψεις όπως είχαμε κάνει στην περίπτωση του ΣΥΣ2 το 2003. Δεν είμαστε στην ίδια φάση. Το κόστος είναι αυτό που είναι λοιπόν, διότι κάτι μάθαμε από τα προηγούμενα λάθη μας. Επίση, συμπεριλαμβάνουν τα πάντα, καλύπτουν τα πάντα. Αυτό είναι ένα ακόμη στοιχείο σημαντικό για τη σημερινή συζήτηση. Μιλάμε για δι, γιατί θέλουμε να καλύψουμε τα πάντα και για το αρχικό σύστημα και από την πλευρά την ευρωπαϊκή αλλά και από την πλευρά των κρατών μελών. Το συνολικό λοιπόν κόστο θα αφορά και την ανάπτυξη και τα χρόνια λειτουργία του συστήματο αυτού βάσει το 2020 που καλύπτει και το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο αλλά θέλουμε να καλύπτονται όλα. Γιατί τώρα 500 δι. Νομίζω ο κύριο Έντσου και κάποιοι άλλοι ε, το επεσήμαναν αυτό και είπαν κάτι και για τη μελέτη αντικτύπου και του τελικού αριθμού που αναφέρονται εκεί. Αυτό το προτείναμε γιατί η διάρκεια, η χρονική διάρκεια που ε, έλαβε υπόψη τη σημαντική αντικτύπου ήταν μεγαλύτερη από ό,τι προβλέπει το πολιτισμό οικονομικό πλαίσιο. Στην μελέτη αντικτύπου η υπόθεση είναι ότι η πρόταση θα εγκριθεί ήδη το 2014 και θα αρχίσει να αναπτύσσεται το σύστημα από το 2015. Τώρα όμω, με το σημερινό μα σχεδιασμό, βλέπουμε ότι η έγκριση, εάν προκύψει, θα προκύψει το 2015 και το 2016 θα αρχίσει να λειτουργεί το σύστημα. Ένα χρόνο λιγότερο λοιπόν. Ω προ την ανάπτυξη και τη λειτουργία και το ανάλογο κόστο. Αυτό εξηγεί και τη διαφορά μεταξύ τη μελέτη αντικτύπου και τα τη στοιχεία και τη σημερινή πρόταση. Επιπλέον, αυτό το υψηλό κόστο ε, δικαιολογείται. Εντάξει, ναι, είναι υψηλό. Όμω, να πω ότι μιλάμε για κόστο το οποίο εκ των υστέρων θα επιτρέψει να κάνουμε οικονομίες, οικονομίες στα κονδύλια που αφιερώνουν, αφοσιώνουν τα κράτη-μέλη τι προσπάθειε διαχείριση των συνόρων του. Και επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για ολοκληρωμένη διαχείριση εδώ. Το αναφέρει και μελέτη εντυπτύπου. Θα σα έλεγα μάλιστα να δείτε και τα παραδείγματα που συνοδεύουν την μελέτη εντεκτύπου και θα καλούσα όλου του βουλευτέ να τα κοιτάξουν, διότι ακριβώ εκεί εξηγείται πώ μακροπρόθεσμα θα κάνουμε απο... ε, οικονομίες, οικονομίες που θα εξισορροπήσουν το αρχικό υψηλό κόστο. Τώρα, εάν μπορεί να υλοποιηθεί αυτό, εάν είναι εφικτό, εντάξει κατάλαβα, Πολύ σύντομα. Μπορεί να υλοποιηθεί. Οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν τα κατάφεραν, μα είπατε. Το σύστημα εισόδου-εξόδου ήταν τελείω διαφορετικό από ό,τι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνοι όμω δεν καταγράφουν την έξοδο. Οπότε δεν μπορούν και να εφαρμόσουν το σύστημα που εμεί προσπαθούμε να εφαρμόσουμε. Και τέλο, η πρόσβαση των διοκτικών αρχών. Να επιστήσω την προσοχή σα στο εξή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και αυτό δεν αναφέρεται στι υποθέσει τη πρόταση, έχει αποδεκτικά στοιχεία που πιστεύουμε δείχνουν ότι θα είναι πολύ υποφελές να έχουν πρόσβαση από την αρχή και οι ιδιοκτικές αρχές στο σύστημα αυτό και την βάση δεδομένων. Ευχαριστώ πολύ. Now the council. Το Συμβούλιο, λίγα λόγια, πριν περάσω στους εισηγητές. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής, σας ευχαριστώ που με την μου δώσατε τη δυνατότητα να παρουσιάσω τις απόψεις του Συμβουλίου γύρω από τη συγκεκριμένη πρόταση. Οι προτάσεις ε, που έγιναν ITPKES και οι οποίες είναι υπό εξέταση ε, εξετάζονται και στα πλαίσια της ομάδας εργασίας ε, της αρμόδιας στο Συμβούλιο η οποία ξεκίνησε να συνεδριάζει κατά τη διάρκεια της Ιρλανδικής Προεδρίας. Δεν θα είναι δυνατόν να καταλήξουμε σε μια συμφωνία βέβαια πάρα πολύ γρήγορα. Οι διαπραγματεύσεις για τις προτάσεις αυτές αποδεικνύονται πάρα πολύ ιδιαίτερα περίπλοκες απαιτείται μια προσεκτική ανάλυση των προτάσεων, του κόστους των προτάσεων και ε, του ωφέλους το οποίο θα προσφέρουν. Τίθενται επίσης και τα, τα θέματα μάλλον της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τα οποία και αυτά πρέπει να αναλυθούν προσεκτικά και σε επίπεδο Συμβουλίου. Θα προσπαθήσουμε πάντως να καταλήξουμε ε, πριν από το τέλος του χρόνου σε κάποια από τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ ε, τους δύο εισηγητές, τον κύριο Έντσιο και την κυρία Ζώμα, για τις προτάσεις τους και θα συνεχίσουμε την ανταλλαγή απόψεων με τις ομάδες εργασίας της αρμόδιας του Συμβουλίου. Η παραδοσιακή συνεργασία ανάμεσα στα δύο όργανα θα συνεχιστεί. Εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να ευχαριστήσω και την ομάδα εργασίας 29 και ε, τους εκπροσώπους των υπολείπων ομάδων εμπειρογνωμόνων. Οι απόψεις τους θα ληφθούν υπόψη. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Θα ακούσουμε τώρα τις ε, τελικές ε, απόψεις των δύο εισηγητών, των εισηγητών μάλλον της κυρίας Ζώμα πρώτα και του κυρίου Έντσιου μετά. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη. Ευχαριστώ τους ε, συναδέλφους ε, για τις απόψεις τους. Θα ήθελα να, να τονίσω ότι ακριβώς γι' αυτό δεν υποβάλαμε ε, έκθεση. Γι' αυτό έχουμε υποβάλει έγγραφα εργασίας για να τα συζητήσουμε μαζί σας. Λίγο περίεργες βρήκα τις κάπως επιθετικές παρεμβάσεις και από τις ε, απαντήσεις βγάζουμε τα συμπεράσματά μας ε, και θα δούμε τι μορφή θα λάβει η έκθεσή μας. Οι ε, επιφυλάξεις που ακούστηκαν εξηγήθηκαν και όλα σε νέα πράγματι το κόστος είναι σοβαρό πρόβλημα και ο συνάδελφος Ένσιο και εγώ βλέπουμε επικριτικά τις ε, δηλώσεις ε, της Κομισιόν ότι το κόστος ε, είναι περιορισμένο. Ξέρουμε τι έχει γίνει σε άλλες περιπτώσεις, γιατί να είναι διαφορετικά τώρα, ωστόσο ο εκπρόσωπος της Κομισιόν είπε ότι έχουν συλλεγεί εμπειρίες από τα συστήματα που είχαμε μέχρι τώρα, ώστε να μπορέσουμε να περιορίσουμε το κόστος και αυτό δεν θα πρέπει να το παραβλέψουμε. Όσον αφορά τη συλλογή βιομετρικών δεδομένων, αυτό είναι πάντα θέμα συζήτησης. Τίθεται λοιπόν το θέμα εάν είναι απαραίτητη η συλλογή τέτοιων στοιχείων και σε τι βαθμό θα πρέπει να πραγματοποιείται. Είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο έχουμε αναρωτηθεί και εμείς. Ε, το θέμα των ε, συνόρων είναι ένα από τα σοβαρότερα. Των χερσαίων συνόρων ε, έχουμε σκεφτεί πώς ε, θα το ε, χειριστούμε. Μπορούμε να έχουμε ένα τέτοιο νέο ηλεκτρονικό σύστημα σε κάθε σημείο εισόδου στα σύνορα. Το έχουμε συζητήσει λοιπόν και αυτό θα ήθελα να τονίσω. Αυτό που είπε και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Ότι δεν ότι το θέμα μας δεν είναι μόνο οι παράνομα διαμένοντες, αυτοί που μένουν πέρα από το διάστημα που δικαιούνται. Αλλά θα ήθελα να πω και το γράφω αυτό και στο έγγραφο εργασίας ότι υπάρχουν συστήματα σε κάποια κράτη-μέλη που προσπαθούν να καταχωρήσουν τις εισόδους και εξόδους σε ταξιδιωτών συλλέγουν ε, αλφαβητικά και αριθμητικά στοιχεία και στόχο ε, έχουν να δώσουν δυνατότητες αρχές επιβολής του νόμου να αποθηκεύουν τέτοια δεδομένα. Και επιπλέον, τα κράτη-μέλη που έχουν τέτοια συστήματα θεωρούν θετικές τις εμπειρίες τους με αυτά, αλλά τα μέλη του Σέγγεν που έχουν τέτοια συστήματα λένε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει κάτι τέτοιο εάν δεν υπάρχει ένα συνολικό ευρωπαϊκό σύστημα για την ανταλλαγή των δεδομένων και νομίζω ότι αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο πρέπει να μας οδηγήσει σε περαιτέρω συζητήσεις. Συνεργάζομαι στενά με τον συνάδελφο Ένσιο, θα συζητήσουμε λοιπόν και το θέμα αυτό. Και θα σκεφτούμε τις συστάσεις, θα υποβάλουμε στην εκθεσή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο παρακαλώ. Καταρχήν ε, να ευχαριστήσω όλους ε, τους ε, συναδέρφους για τις παρεμβάσεις τους, τις ιδέες τους. Θα ληφθούν όλες οι παρατηρήσεις υπόψη στο σχέδιο της έκθεσης. Δεν θα επαναλάβω αυτά που ήδη υπόθηκαν. Ένα πράγμα θα ήθελα να τονίσω ότι όλα τα έγγραφα από την Κομισιόν ε, για του, τα εφή e συστήματα ταξιδιωτών ε, έχουν ε, γίνει χωρίς αξιολόγηση της αναγκαιότητας και αναλογικότητας των νέων μέτρων με βάση τα, τα δεδομένα. Δεν μας επιτρέπει η πρόταση αυτή να επικεντρωθούμε στο πρόβλημα ε, και τις ε, πιθανές λύσεις. Στις ε, μελέτες αντικτύπου της Κομισιόν υπάρχουν πράγματα τα οποία αμφισβητούνται κάπως στις στη μελέτη επιπτώσεων του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να ζητήσω μια δεύτερη θεσμική εξέταση των, του αντικτύπου της πρότασης ε, για τα ευφυή e συστήματα ταξίδιωτών. Οι ε, ανησυχίες ε, που εκφράστηκαν για τα δύο αρχικά πακέτα νομίζω ότι αιτιολογούν ένα τέτοιο βήμα. Χαίρομαι που ήταν τόσο καλή αυτή η συζήτηση και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Λοιπόν, είχαμε μια εξαντλητική συζήτηση και τώρα έχουμε μείνει πίσω δυστυχώς. Έχουμε θέμα χρόνου σοβαρό και θα περάσουμε στο επόμενο θέμα αμέσως. Το 11 θα ακούσουμε την παρουσίαση των εμπειρογνωμόνων από το ECTR. Είναι, ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Ανοχή και τη Συμφιλίωση δημιουργήθηκε το 2008 από τον Αλεξανδάρ Κβανιεύσκη, τότε πρόεδρο της Πολωνίας και τον Μωσέ Καντό, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού ε, Ισραηλιτικού Κογκρέσου. Στόχος είναι η καταπολέμηση του ρατσισμού, του αντισημιτισμού και της ξενοφοβίας. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν και πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές η διάσκεψη των Προέδρων ζήτησε από την Επιτροπή μας να συναντηθούμε με εκπροσώπους του ECTR και γι' αυτό σήμερα καλωσορίζουμε τους εκπροσώπους τους ε, ε, εκπροσώπους της Επιτροπής Νομικών Εμπειρογνωμόνων του ECTR. Έχω εδώ κάποιους, ε, κάποια από τα ονόματα των προσκεκλημένων. Παρακαλώ αν μπορείτε 5, ε, με 7 λεπτά ο καθένας έτσι ώστε να παραμείνει λίγος χρόνος για την ε, συζήτηση. Θα δώσω πρώτο τον λόγο στον καθηγητή Γιωράμ Ντίνσταϊν ο οποίος είναι τέος πρόεδρος του Πανεπιστημίου του Τελαβίβ, είναι πρόεδρος ε, της, Ένωσης, της Ισραηλινής Ένωσης Διεθνούς Δικαίου και μετά θα δώσω τον λόγο στον κύριο Ούγκο Τζενέζιο, ο οποίος είναι τέος δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου και συνειδητής ε, του ε, Ινστιτούτου του Σαν Ρέμο για το Ανθρωπιστικό Δίκαιο και θα έχουμε επίσης και τον κύριο Μπιλ που είναι νομικός εμπειρογνώμων από πλευράς του ECTR. Λοιπόν θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Μπίλ. Έτσι θέλετε. Ο κύριος Μπίλ λοιπόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας και ευχαριστώ και την Επιτροπή Λίμπε. Λέμε, λέγομαι Γκενάουις Μπίλ, είμαι γραμματέας της ε, Επιτροπής μας, του Συμβουλίου μας που δημιουργήθηκε το 2008 μετά από απόφαση κοινή του κύριου Κβασνιεύσκη και του κύριου Καντόρ, αλλά συμμετέχουν και άλλες προσωπικότητες, τέως πρόεδροι, τέως πρωθυπουργοί, όπως ο Χωσέ Μαρία Σνάρ, ο Πέρσμαν, ο, ε, από τη Λετωνία, η Ρίτα Ζίσμουθ από την Γερμανία, ο Γιώργος Βασιλείου από την Κύπρο, και τα λοιπά. Υπάρχουν πάρα πολλές προσωπικότητες οι οποίες με τη ζωή τους και τις πολιτικές τους δραστηριότητες έχουν προωθήσει την ιδέα της συμφιλίωσης και της ανοχής. Ήταν μέλος μας και ο Βακλά βέβαια. Κυρίες και κύριοι, το σχέδιο αυτό το οποίο προσπαθούμε να προωθήσουμε ξεκίνησε το 2011 τρία χρόνια μετά την έναρξη ε, της, ε, της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη και ανάμεσα σε πάρα πολλές δηλώσεις ε, Ευρωπαίων πολιτικών σχετικά με την αποτυχία των πολυμερών διπλωματικών σχέσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταπολέμηση του ρατσισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο ΑΣΕ, έχουν παρουσιάσει εκθέσεις και έχουν προειδοποιήσει για την αύξηση της ξενοφοβίας και των φαινομένων ρατσισμού στην Ευρώπη. Εκείνη την εποχή οργανώσαμε μια διεθνή διάσκεψη για τη συμφιλίωση στα Βαλκάνια το 11 και κατά τη διάρκεια αυτής της διάσκεψης αποφασίσαμε να ζητήσουμε τη γνώμη μια σειρά νομικών εμπειρογνωμόνων γνωστών Ευρωπαίων οι οποίοι θα μας παρουσίασαν τη νομική κατάσταση των πραγμάτων σε διάφορες χώρες της Ένωσης και θα προσπαθούσαν όχι μόνο να δούνε ποιος είναι ο νομικός ορισμός της ανοχής, αλλά της έννοιας ανοχή, αλλά και ε, ποιες είναι οι νομικές ρυθμίσεις σε θέματα συγκεκριμένα όπως η κλειτοριδοεκτομή, όπως η μπουρκα, και τα λοιπά αντίστοιχα τέτοιου είδους θέματα και άλλα πρακτικά επιμέρους θέματα τα οποία είχαν συζητηθεί εν πολλής ε, ε, στα πλαίσια των ενδιαφερόντων της κοινή γνώμης. Εμείς ε, καταλήξαμε σε συγκεκριμένα έγγραφα, τα παρουσιάσαμε το 2012, εμείς δώσαμε και στον Μπόρι Τάντιτς το βραβείο για την προώθηση της ε, της ανοχής και της συμφιλίωσης των λαών. Από τότε συζητήσαμε το θέμα αυτό και με το Συμβούλιο της Ευρώπης τα πλαίσια της Επιτροπής που έχει δημιουργήσει για την καταπολέμηση του ρατσισμού με το Συμβούλιο για τον Σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Βαρσοβία και μιας και προβλέπεται το θέμα αυτό να γίνει δεκτό ε, και από τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Έχουμε επισκεφθεί αρκετές πρωτεύουσες, έχουμε πάει στη Ρουμανία, στη Ρουμανία έχουμε προχωρήσει και θα συζητηθεί στο κοινοβούλιο και θα γίνει δεκτό σύντομα. Έχουμε επίσης προετοιμάσει μια αντίστοιχη διάσκεψη και παρουσίαση στη Βουδαπέστη, ε, όπως επίσης και στην Πράγα και περιμένουμε να οργανώσουμε συναντήσεις και σε άλλες χώρες όπως το Βερολίνο, το Παρίσι και η Μαδρίτη. Δεν θα μακρηγορήσω, θα δώσω το λόγο στον καθηγητή Ντίνσταϊν, ο οποίος είναι πρόεδρος της ομάδας νομικών εμπειρογνωμόνων και ο οποίος θα παρουσιάσει το περιεχόμενο της συγκεκριμένης πρότασης. The second floor goes to Mr. The chair. Το λόγο τώρα ο κύριος Ντίνσταϊν, ο πρόεδρος της Επιτροπής για την Ανοχή στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Μετά από την εισαγωγή αυτή θα ήθελα να προχωρήσω κατευθείαν στην ουσία. Επιτρέψτε μου καταρχήν ε, να αναφερθώ στις ε, επανειλημμένες ε, δεσμεύσεις για ανοχή και στην Ευρώπη και αλλού. Αλλά η δέσμευση αυτή είναι γενική, δεν έχει μορφή το θέμα είναι ότι κανένας δεν θεωρεί τον εαυτό του ε, ως μυσαλόδοξο. Εγώ τουλάχιστον ε, δεν έχω συναντήσει κανένα τέτοιον άνθρωπο στη ζωή μου. Ωστόσο, κανένας ε, δεν γνωρίζει τι ακριβώς ε, είναι η ανοχή. Και το περίεργο είναι ότι καμία συνθήκη δεν καθορίζει τον όρο αυτό ούτε στην Ευρώπη ούτε σε παγκόσμιο επίπεδο. και όλοι επικεντρώνονται σε διαφορετικό θέμα που είναι οι διακρίσεις στο Στρασβούργο. Ο κόσμος εξεπλάγει ότι ε, η ανοχή είναι θέμα ε, ε, ξεχωριστό από τις από τις διακρίσεις και έπρεπε να δείξουμε ότι κάποιος μπορεί να είναι μυσαλόδοξος χωρίς να κάνει διακρίσεις. Γιατί λοιπόν υπάρχει αυτή η τάση αποφυγή του θέματος αυτού. Θα μπορούσαν να δοθούν πολλές απαντήσεις. Ε, εγώ βεβαίω δεν είμαι, αλλά υποψιάζομαι ότι συμβαίνει επειδή ε, πολλοί ε, κόσμος ε, που ασχολείται με τις πολιτικές ελευθερίες είναι μπερδεμένος διότι ε, από τη μία, ναι φυσικά όλοι είμαστε υπέρ τη ανοχή, ωστόσο όλοι γνωρίζουμε λόγω των γεγονότων ε, στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχουν ε, μέρη και εποχές ε, όπου νιώθει κανείς πολύ βαθιά ότι όσο και να είναι υπέρ της ανοχής ε, κάπου θα πρέπει να υπάρχει και κάποια εξαίρεση. Δεν μπορεί να θέλει να το πει κανείς ανοιχτά, οπότε το αποφεύγει. και ε, ζητώ συγγνώμη, ε, δεν εννοώ εσείς εσείς, ε, μιλώ για όλους τους ανθρώπους. η, η Vox Populi, η φωνή του λαού στις ευρωπαϊκές χώρες αλλάζει συνέχεια και νομίζω ότι όλοι γνωρίζετε ότι δυστυχώς ε, υπάρχουν τάσεις προς τις λάθος κατευθύνσεις στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης ε, σήμερα. Και για το λόγο αυτό πιστεύουμε ότι δεν μας παίρνει να ε, αποφύγουμε το ζήτημα του αντίον, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και αυτό θα πρέπει να γίνει με την εθνική νομοθεσία εθνική νομοθεσία η οποία θα δημιουργήσει σε κάθε χώρα ξεχωριστά ε, έναν τύπο που θα βασίζεται σε ε, κοινό παρονομαστή, τον οποίο πολύ ευχαριστώ να παράσχουμε εμείς. Αυτό προσπαθήσαμε λοιπόν να κάνουμε. Το κείμενο που έχουμε εκπονήσει και που έχει διανεμηθεί, κάποιοι από εσά μπορεί να το έχουν διαβάσει, ελπίζω ότι θα το έχετε διαβάσει, ε, είναι απλά ένα πλαίσιο δεν είναι οριστικό, δεν είναι μία πρόταση από την οποία θα πρέπει να δεχτείτε ή όλα ή τίποτα. Του αντίον πιστεύουμε ότι θα πρέπει να μπορεί να προσαρμόζεται στις ανάγκες ε, της κάθε χώρες. Ε, δηλαδή, ε, σε κάποιες χώρες η ολα η τιποτα του μπορεί να έχει κάποιος διαφορετική μορφή αρκεί να προσαρμοζεται στις αναγκες της καθε χωρες δηλαδη σε καποιες χωρες η νομοθεσια μπορει να εχει καποιες διαφορετικη μορφη αρκει να εχει τον κοινό παρονομαστή. Και ποιος είναι αυτός ο κοινός παρονομαστής. Στην ουσία του είναι ότι υπάρχει μια διχοτομία, υπάρχει το δικαίωμα του να είναι κανείς διαφορετικός ε, και από την άλλη ε, σε κάθε χώρα υπάρχει μια κοινωνία με ε, ειδική ταυτότητα και τα δύο αυτά θα πρέπει να ταιριάξουν μεταξύ τους και ακριβώς αυτή είναι η πρόκληση πώς μπορούμε να έχουμε ε, μία ενιαία κοινωνία χωρίς αφομοίωση των διαφόρων ομάδων και από την άλλη πώς μπορούμε να έχουμε επικοινομορφία χωρίς διάλυση του κράτους, ε, της χώρας. Ε, θέλουμε επικοινομορφία χωρίς διάλυση και αποτέλεσμα... Το αποτέλεσμα είναι η συνύπαρξη που αποτελεί συμβιβασμό και πιστεύουμε ότι η ποικιλομορφία με την συνύπαρξη δεν θα πρέπει να είναι πυρηταποθήκη, θα πρέπει να είναι η, η κόλλα που ενώνει την κοινωνία. Υπάρχουν λοιπόν εννέα τμήματα στο εγγραφό μας και θα ήθελα να σας τα παρουσιάσω πολύ σύντομα. Το ε, πρώτο τμήμα ξεκινάει με τέσσερις ορισμούς. Ε, κανένας ε, από τους ορισμούς αυτούς ε, δεν μπορεί να σας φαίνεται ιδιαίτερα ιδιαίτερα πρωτότυπος, αλλά είναι. Έχουμε χρησιμοποιήσει στοιχεία από άλλα κείμενα, αυτό το κάναμε ε, ηθελημένα, αλλά πουθενά δεν θα βρείτε τους τέσσερις αυτούς ορισμούς με τη μορφή που έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε λοιπόν ε, την ε, ανοχή, την ομάδα, την ε, ομαδική συκοφαντία και τα εγκλήματα μίσους. Την ανοχή λοιπόν, όσον αφορά την ανοχή, ακούσατε τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να έχουμε ε, συνδυασμό της επικοινομορφίας αλλά και μιας ενιαίας κοινωνίας. Όσον αφορά τις ομάδες, εδώ ακολουθήσαμε την ε, παραδοσιακή αναφορά σε ε, πολιτιστικές και φιλετικές ρίζες, αλλά εθνοτικές, αλλά ακολουθώντας και πιο πρόσφατες εξελίξεις έχουμε συμπεριλάβει και και άλλα στοιχεία ε, όπως είναι η ταυτότητα του φύλου και, η ε, σεξουαλική, ε, και ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Ενδεχομένως στο μέλλον να συμπεριληφθούν και άλλα στοιχεία. Πάντως τα στοιχεία αυτά που έχουμε εδώ είναι σημαντικά. Όσον αφορά λοιπόν την ομαδική δυσφήμιση, αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι ε, συχνά ο κόσμος πιστεύει ότι ε, κάτι θα πρέπει να απαγορεύεται μόνο όταν αποτελεί παρακίνηση για βίαιες πράξεις. Ε, προφανώς αυτό είναι δεδομένο, αλλά πέρα από αυτό ε, ακόμα και απλά η ε, συκοφαντική δυσφήμιση ή ε, η γελιοποίηση θα πρέπει να απαγορεύεται. Όπως το να λέμε ότι όλοι οι τσιγκάνοι είναι κλέφτες, όπως και τα εγκλήματα μίσους, τα οποία παντού ορίζονται, αλλά εμείς έχουμε τον πιο απλό ορισμό. Λέμε ότι το έγκλημα μίσους είναι ένα απλό έγκλημα, το οποίο όμως γίνεται ιδιαίτερο διότι συνδέεται με με, ε, με μια συγκεκριμένη ομάδα. Δηλαδή, μπορεί να μιλάμε για φόνο, για επίθεση, για ε, ε, έγκλημα όμως το οποίο πραγματοποιείται επειδή το θύμα ανήκει σε μια συγκεκριμένη ομάδα. Αυτό λοιπόν είναι το θύμα 1. Το τμήμα 2 αναφέρεται στην ξενοφοβία, τον αντισημιτισμό, τον ε, αντιφεμινισμό ε, και, ε, και τις διακρίσεις εις βάρος ομοφιλοφίλων. Το τμήμα 3 αναφέρεται στα σχετικά ανθρώπινα δικαιώματα και το βασικό στοιχείο που προσθέτουμε εδώ πέρα ε, είναι ότι θα πρέπει να δούμε το θέμα αυτό όχι μόνο ε, εγκάρσια, να δούμε δηλαδή τις ε, σχέ... όχι να, μην το δούμε μόνο κάθετα, δηλαδή τις σχέσεις κράτους και ατόμου, αλλά θα πρέπει να δούμε και τις σχέσεις μεταξύ των διαφορών ομάδων. οι ομάδες θα πρέπει να σέβονται η μία την άλλη. οι εκπρόσωποι ομάδων υποστηρίζουν ότι χρειάζονται προστασία ιδιαίτερη μεταχείριση κλπ. Όσον αφορά όμως άλλες ομάδες ξαφνικά σωπαίνουν. Ε, το τμήμα 4 ε, έχει να κάνει με τους ε, περιορισμούς διότι θέλουμε να πούμε στους ανθρώπους που ασχολούνται με τις πολιτικές ομάδες είναι ότι η ανοχή δεν μπορεί να ε, είναι χωρίς όρια. Δεν μπορεί κανείς να δείχνει ανοχή απέναντι στους ε, ε εάν δηλαδή μία ομάδα ε, είναι κατά της ανοχής, είναι μυσαλόδοξη, τότε δεν της αξίζει να τις φορόμαστε κι εμείς με τέτοιο τρόπο. Και αναφερόμαστε για παράδειγμα ε, αναφερόμαστε για παράδειγμα στον ε, ακροτηριασμό των ε, γυναικών ή άλλες τέτοιες πρακτικές. Εκεί δεν θα πρέπει να υπάρχει ανοχή. Η ανοχή γενικά όμως θα πρέπει να είναι αμοιβαία. Και το τμήμα 5 ασχολείται με τους μετανάστες, το οποίο ε, είναι ίσως το πιο καυτό θέμα σήμερα στην Ευρώπη. Και εμείς ε, προτείνουμε από τη μία να ε, είμαστε ανοιχτικοί απέναντι όχι μόνο σε παλαιές ομάδες, αλλά και απέναντι σε νέες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων μεταναστών. Και από την άλλη, αν έχουμε μετανάστες που δεν σέβονται την αρχή συνύπαρξης εντός μιας κοινωνίας, τότε εφόσον ε, το άτομο αυτό δεν είναι πολίτης ε, της ε, κοινωνίας, τότε η κοινωνία είναι, έχει ένα πλεονέκτημα διότι μπορεί να πει ότι έχετε απεπολύσει το δικαίωμα να παραμείνετε στη χώρα. Έναν πολίτη δεν μπορούν να τον απελάσουν από τη χώρα, αλλά έναν μη πολίτη της χώρας μπορούν. Αυτό λοιπόν το θέμα είναι πολύ λεπτό, είναι μια πολύ απλή λύση σε ένα καυτό ερώτημα. Το τμήμα 6 έχει να κάνει με την εφαρμογή. Εδώ λοιπόν έχουμε μία νέα πρόταση. Ε, όχι μόνο να έχουμε κυβερνητικές ε, διοικητικέ επιτροπές ε, που να εποπτεύουν το θέμα αυτό. Αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο φυσικό και αυτονόητο. Συμβαίνει σε πολλές χώρες αλλά να έχουμε μία εξωτερική ε, ομάδα, να έχουμε ε, μία εθνική ανεξάρτητη ε, επιτροπή παρακολούθησης θεμάτων ανοχής. Θα πρέπει λοιπόν αυτός ο φορέας να έχει αρμοδιότητες να παρακολουθεί την κατάσταση, να υποβάλει προτάσεις και θα επανέλθω στο θέμα αυτό σύντομα. Το τμήμα 7 έχει να κάνει με τις ποινικέ κυρώσεις. Θέματα ε, συγκοφάντηση συγκοφάντησης ή εγκλημάτων μίσους είναι πολύ σημαντικά. Ε, ασχολούμαστε και με το θέμα των ε, ανηλίκων κλπ. Το τμήμα 8 ε, ασχολείται με την εκπαίδευση. Εδώ έχουμε την ουσία του όλου θέματος, διότι η εκπαίδευση είναι απολύτως απαραίτητη και είναι απαραίτητη ε, από την κούνια μέχρι τον τάφο. Θα πρέπει δηλαδή να καλύπτουμε εδώ την εκπαίδευση και των νέων και των ενηλίκων. Ε, και επίσης ε, θέμα είναι πώς θα εκπαιδεύσουμε τους εκπαιδευτές. ακόμα και δικαστές, σίγουρα τους νομικούς, ε, καθώς και τους στρατιωτικούς, την αστυνομία κλπ. Δεν είναι πολύ απλό το θέμα, ε, πρέπει να γίνει όμως και μπορεί να γίνει κατά τη γνώμη μας. Τέλος, το τμήμα 9 ασχολείται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αναπτύξουν ε, ηθικούς κώδικες. Δεν θέλουμε όμως ε, κυβερνητικό έλεγχο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Θα πρέπει λοιπόν να υποπτεύονται μόνο τους. Έχουμε και το θέμα του διαδικτύου, το οποίο έχουμε αποφύγει θελημένα, διότι Συζητείτε πώς μπορεί κανείς ε, να εποπτεύει το διαδίκτυο. Σκεφτήκαμε λοιπόν να περιμένουμε ε, όσον αφορά το θέμα αυτό. Συνοψίζοντας, η Ευρώπη δεν ε, μπορεί να αποφύγει το ζήτημα, πρέπει να το αντιμετωπίσει. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Πιστεύουμε ότι εσείς ως Επιτροπή αλλά και ως μεμονωμένοι Ευρωβουλευτές μπορείτε να μας βοηθήσετε ώστε να περάσει τέτοια εθνική νομοθεσία και θα χαιρόμασταν αν η ΛΥΜΠΕ μπορεί να εγκρίνει την ιδέα του προγράμματος αυτού. Ε, και πάλι δεν μας ενδιαφέρουν εδώ οι λεπτομέρειες ε, που μπορείτε να δεχτείτε ή όχι. μας ενδιαφέρει η κατεύθυνση που ακολουθούμε και όχι οι λεπτομέρειες. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Make πάρα πολύ σύντομα σχόλια για να μείνουν και λίγα λεπτά για τα μέλη μας να πάρουν το λόγο. Ο κύριος Βενέτσιο, δικαστής από την Ιταλία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Όμως οι παρουσιάσεις των συναδέλφων νομίζω ήταν αρκετά διεξοδικέ και πλήρε. Ανέφερε ο συνάδελφο όσα ήθελα να πω στην επιτροπή σα. Απλώ να σημειώσω ότι η δική μα ομάδα εμπειρογνωμόνων συμπεριλαμβάνει και τρει συναδέλφου οι οποίοι δεν μπόρεσαν να παραστούν σήμερα στη συνεδρίαση. Ο καθηγητή Ράιν Μιλέσον από την Εστονία, ο καθηγητή Ντάνιελ Τούρερ από την Ελβετία και ο κύριος Λούντιγκε Βόλθαμ από τη Γερμανία. Να σας αφήσω πραγματικά το πεδίο ελεύθερο για να συζητήσετε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ για τη σύντομη αυτή σας παρέμβαση. Πολύ καλό αυτό. Οπότε μπορούμε να ακούσουμε τώρα και τους ε, βουλευτές μας. Κυρία Σίπελ, μπορείτε να ξεκινήσετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω το ECTR για τη δουλειά που έχει κάνει. Πρέπει όμως ε, να πω επίσης ότι δεν με πείθει απολύτως το αποτέλεσμα. Καταρχήν αναφέρθηκε ότι μιλάμε πολύ για διακρίσεις, δεν μιλάμε πολύ όμως για την ανοχή. Οι ίδιοι όμως ε, στην εισαγωγή του γράφου τους λένε ότι Ανοχή είναι το αντίθετο της, ε, ε, των διακρίσεων. Οι διακρίσεις είναι μια συγκεκριμένη πράξη κατά της οποίας ε, μπορώ κάτι να κάνω. Για παράδειγμα, δεν σου δίνω δουλειά επειδή, δεν έχεις, επειδή είσαι ξένος. Απέναντι σε αυτή την πράξη μπορώ κάτι να κάνω, αλλά η μυσαλλοδοξία είναι κάπως πιο δύσκολο θέμα και σε κάποια θέματα νομίζω ότι θα πρέπει να ενεργήσουμε περισσότερο πολιτικά. Αναφερθήκατε σε μυσαλόδοξη συμπεριφορά και ε, στην, ε, στον μη σεβασμό των άλλων, ε, αλλά αυτό δεν είναι το θέμα. Τι θα κάνω με τους δικούς μου πολίτες που, επιδεικνύουν τέτοια συμπεριφορά και γι' αυτό το θέμα της ε, απέλασης ε, δεν μας βοηθάει. Θα πρέπει ως κοινωνία να ασχοληθούμε με τέτοιες συμπεριφορές ε, και θα πρέπει η δημοκρατία να ενισχυθεί ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν τέτοια θέματα. Και επικριτικά βλέπω επίσης ε, το θέμα θα πρέπει να υπάρχει μάθημα ε, διδασκαλίας ε, για την άνοχη. Η ανοχή για μένα είναι μια στάση απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Δεν μπορώ να το διδάξω αυτό ή να το μάθω όπως την προπαίδεια. Και Σημαντικό είναι αυτό που γίνεται σε κάποια σχολεία. Από κάποια ε, μέρη του μαθήματος των θρησκευτικών ε, ασχολείται με το θέμα αυτό. Αλλά μάθημα ανοχής βρίσκω ότι μάλλον είναι προβληματικό ως θέμα. Κυρία Ζήπελ, σας παρακαλώ. Και μία τελευταία πρόταση, κύριε Πρόεδρε, για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ε, πιστεύω ότι ε, τις τελευταίες εβδομάδες ε, και μήνες είχαμε πολλές συζητήσεις ε, για την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το να υπαγορεύουμε λοιπόν συγκεκριμένα ποσοστά του χρόνου τους που θα πρέπει να αφιερώσουν σε κάποιες ιδέες βρίσκω ότι είναι προβληματικό θέμα. Έχω λοιπόν ερωτήσεις σχετικά με το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε με τις προτάσεις ε, που μας έχουν υποβληθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. κύριος Μπρόγκς, παρακαλώ όμως προσπαθείτε, προσπαθείτε σε ένα δίλεπτο να ολοκληρώνετε, διότι έχουμε και την συνεδρία των συντονιστών αμέσως μετά. Πρέπει να γίνει και αυτή. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, είναι χαρακτηριστικό του, τη βλέπουμε και στην ε, τηλεόραση, ότι δεν αναγνωρίζονται πάντοτε όσα αναφέρονται ηρωνικά ή με τρόπο και βλέπουμε επεισόδια φυλάκισης ή μη καταπολέμησης ε, ρατσιστικών φαινομένων. Το... Η χρήση υπερβολικών όρων με μία απόλυτη κατανόηση του ακριβούς νοήματός τους από ανθρώπους που θέλουν σε αυτός τους ε, πανεπιστημιακούς είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Η ξενοφοβία, ο φόβος των αεροδαπών είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό και ε, ε, διαδεδομένο πλέον στις μέρες μας. Το ίδιο όμως και η δίωξη για τέτοια θέματα. Το να δημιουργούμε μια πανεπιστημιακή κατάρτιση για το θέμα αυτό, μια ακαδημαϊκή προσέγγιση για τα φαινόμενα αυτού του τύπου, δείχνει πόσο λανθασμένη είναι μια τέτοια οπτική γωνία. Η επιλογή των λέξεων πολλές φορές μας λέει περισσότερα για τις λέξεις τις ίδιες από ό,τι για τους ανθρώπους τους ίδιους και το πώς τις χρησιμοποιούν. Οι λέξεις είναι αυτές που μισούν ε, τους ε, ανθρώπους, όχι οι άνθρωποι. Βλέπουμε τι προβλήματα προκαλούν τα λόγια λόγια στι Ηνωμένες Πολιτείες. Χάνουν πολλές φορές το ακριβέ τους νόημα και ο στόχο τους δεν είναι να σημάνουν κάτι, αλλά να βγάλουν τους ανθρώπους από την ε, ορθολογιστική τους προσέγγιση και να τους προκαλέσουν παράλογες συμπεριφορέ. Η παρότρινση σε μίσος κατά ενός κατηγορουμένου ήταν κάτι που είδαμε πρόσφατα. ή σωματικές επιθέσεις κατά εθνικών μειονοτήτων. Αυτό είναι κάτι που λένε και περισσότερο σπανίζει. Όμως όλο ένα και περισσότερο υπάρχει παρότρινση σε πράξεις μίσους, ιδίες συμπεριφορές ε, και από ανθρώπους που μάλιστα εκφράζουν ε, την ακαδημαϊκή τους απλώς άποψη. Νομίζω ότι αυτό απλώς ζήσαμε σήμερα το πρωί. Ευχαριστούμε, ο κύριος Κλής. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, έχω πολλούς ενδιασμούς και εγώ για αυτή την πρόταση. Θεωρώ ότι είμαι ένας άνθρωπος ε, ανεκτικός. Ε, κανείς δεν μπορεί να μου το αμφισβητήσει αυτό. Ε, και κανείς βεβαίως δεν μπορεί να πει ότι είναι κάτι κακό η ανοχή, η ευγένεια, οι καλοί τρόποι, αλλά δεν ξέρω αν είναι και δημόσιο θέμα, ε, αν μπορούμε να επιβάλλουμε κανόνες, να υιοθετήσουμε νομικές διαδικασίες ή νομοθετικές προβλέψεις. Εδώ είναι λιγάκι σαν να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε δύο φαινόμενα που είναι η, ίδια όψη, η άλλη όψη του ίδιου Από τη μια δηλαδή έχουμε ε, την ξενοφοβία με νομίζω κατά την ταπεινή μου άποψη λύσεις που καλύπτουν τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν έχουμε πάει αρκετά μακριά ως προς το ότι πρόκειται πραγματικά για μια προσπάθεια στέρησης της ελευθερίας, κάτι που αποτελεί και θεμελιώδες δικαίωμα. Και αυτό ακριβώς είναι και το πρόβλημά μου με το συγκεκριμένο κείμενο. Είναι σαν να ε, ασκούμε λογοκρισία και Νομίζω όταν ε, μιλούμε για κανόνες, για ε, τρόπους συμπεριφοράς που επιβάλλονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης λόγου χάρη, ε, αρχίζει το πράγμα να δυσκολεύει. Μπορούμε να προωθήσουμε την ανοχή, την ανεκτικότητα. Μα η ανεκτικότητα και η ανοχή είναι ζήτημα του καθενός. Πρέπει να δούμε και τι λέει, η λογοτεχνία, τι ε, κυκλοφορεί στην τέχνη. Τον επιβάλλουμε τώρα μια τέτοια συμπεριφορά και μάλιστα με ένδικα μέσα που να την ε, τιμωρούν εφόσον ξεπερνά κάποια όρια, αυτό βρίσκονται είναι τελείω παράλογο. Νομίζω λοιπόν ότι το κείμενο που εξετάζουμε είναι τελείω προβληματικό γιατί φαίνεται να μην αναγνωρίζετε του κινδύνου των όσων εξακέλετε. και ενθαρρύνεται. Λέτε όχι, δεν στοχεύουμε την ελευθερία της έκφρασης, αλλά τα πρακτικά της αποτελέσματα. Μα αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ελέγξει κανείς. Όντως επίσης πολύ δυσκολευόμαστε με τη μετανάστευση στην Ευρώπη. Αλλά το να πούμε ότι κάποιοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ε, υπερασπίζονται την ποικιλομορφία, την πολιτιστική ποικιλομορφία, είναι ένα πράγμα. Κάποιο όμω είπε ότι η κυκλομορφία αυτή είναι αποτυχημένη προσπάθεια και ότι δεν έχει κανένα νόημα. Αλήθεια είναι και αυτό. Δεν είναι αρκεί να λέμε ότι η μαζική λαθρομετανάστευση προσφέρει. Μάλλον ότι η λαθρομετανάστευση έχει ξεπεράσει τα όρια και ότι η κυκλομορφία δεν συνδυάζεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε ρατσιστέ. Ευχαριστούμε ο κύριο Γκρίφιν. Ευχαριστώ Αναφέρεται στην ε, παιδεία, στην εκπαίδευση, αλλά όταν μιλάμε για εκπαίδευση πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη πρόταση, το θέμα είναι αντιπαράθεσης ανάμεσα στις γνώμες και τα δόγματα από ένα απομονωμένο κέντρο αριστερό καθεστώς το οποίο ε, είναι εναντίον ε, της μαζικής, ε, είναι εναντίον της κοινής γνώμης και η οποία με τη σειρά της είναι εναντίον της μαζικής μετανάστευσης. Λέει εδώ ότι πραγματικά παροδία του 1984 του βιβλίου αναφέρεται στην χρήση των δημοσίων, του δημοσίου χρήματος για να διώκονται αυτοί οι οποίοι εκφράζουν την άποψη της καταπιεσμένης, καταπιεσμένης πλειοψηφίας. Χρήση των φορολογουμένων και του χρήματος των φορολογουμένων για να καταστέλλεται η άποψη των ιδίων των φορολογουμένων. Πραγματικά βλέπετε εδώ μια εικόνα με τον Άλεξ. Ο Άλεξ είναι από το Clockwork Orange το κουρδιστό πορτοκάλι του Κιούμπρεκ με τη μουσική της Ενάτης Συμφωνίας. Αυτό θα γίνουμε, κουρδιστό πορτοκάλι θα γίνουμε, ε, γελί αλλά και φρικτή ταυτόχρονα μέσω όλων αυτών των απαγορεύσεων ε, και ένα πρόγραμμα σαν το δικό σας το οποίο στην ουσία δημιουργεί μειονότητες μέσω της πλειοψηφίας. Εσείς που προέρχεστε από την εβραϊκή κοινότητα Ξέρετε ότι ταυτίζεστε με το κράτος του Ισραήλ που καταπιέζει τους Παλαιστινίους με ναζιστικό τρόπο. Εσείς κάνετε μία πρόταση γενοκτονική, μία πρόταση που πρέπει να απορριφθεί, μία πρόταση η οποία δεν θα πρέπει να εμποδίσει ε, την, την εικόνα που έχουμε μερικές φορές για τη σύγχυση των ενιών. Ευχαριστώ Πρόεδρε τίποτα καινούριο σε σχέση με τα όσα άκουσα από τους συναδέλφους. Δηλαδή, το τελευταίο 48 ώρο λάβαμε ένα σωρό ε, ειδοποίησεις και επιστολές, κυρίως από τον Αμένο Βασίλειο, που χρησιμοποιούν ακριβώς την ίδια γλώσσα και το ίδιο και τα ίδια παραδείγματα. Πέραν αυτού όμως, και παρόλο που διαφωνώ απολύτως μαζί τους, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είμαστε μάλλον πολύ προσεκτικοί. Όταν νομοθετούμε για τέτοιου ζητήματα στη δική μου τη χώρα, τη Ρουμανία, Υπάρχει νομοθεσία κατά τη διακριτική μεταχείριση και υπάρχει και αρμόδιο οργανισμό που μελετά το φαινόμενο. Θεωρούμε ότι η διακριτική μεταχείριση υπάρχει και το θεωρούμε δεδομένο αυτό. Όμω η εμπειρία των τελευταίων ετών δείχνει ότι συνήθω όλα αυτά ε, τα φαινόμενα αφορούσαν λόγια εκφράσεις που τιμωρούνται από όλες τις αρμόδιες αρχές και από το δικό μας οργανισμό. Βεβαίω ξέρουμε ότι ο διάβολος κρύβεται στι λεπτομέρειες όπως λέει αυτή η έκφραση, και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το πώ νομοθετούμε. Εδώ μιλάμε για μια οδηγία. Μπορεί να υλοποιηθεί από τα κάτι μελη θα πρέπει μάλλον να υλοποιηθεί από τα κάτι μελη εκ των υστέρων. Τι είδου εναρμονισμένη Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουμε. Το γεγονός ότι συζητούμε σήμερα την έκθεση αυτή, νομίζω, είναι πολύ καλό στοιχείο. Διότι ζούμε σε έναν κόσμο όπου πραγματικά μπορούμε να συμπεριφερόμαστε ανάλογα με κάποια βασικά όρια και κάποια αντίληψη του σεβασμού προς τον άλλο η ανοχή και η ανεκτικότητα είναι κάτι που δεν με βρίσκει τελείω σύμφωνο. Πιστεύω ότι υπερέχει ο σεβασμός προς τον άλλο και η ε, ποικιλία. Δεν είναι βεβαίως κάτι που κληρονομεί κανείς γενετικά η ανεκτικότητα και ανοχή. Είναι κάτι που το κερδίζει με την ε, παιδεία και την καλλιέργεια. Από την οικογένειά του, από την κοινωνία, στο σχολείο, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βεβαίως αυτό θα πρέπει να είναι νομίζω γνώμονάς μας και προς αυτή την κατεύθυνση να οδεύσουμε. Και νομίζω ότι ξεκινούμε ένα πολύ μακρύ ταξίδι εφόσον θέλουμε να συζητήσουμε ένα τέτοιο θέμα. Ευχαριστώ. κάποιος συνάδελφος που θα ήθελε για μια, ένα λεπτό μια παρατήρηση, κύριε Μπέκερ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα απλά να τονίσω πόσο χρήσιμη είναι κατά τη γνώμη μου αυτή η πρωτοβουλία τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι υπάρχει αυξηνόμενος αριθμός ε, ρατσιστικών συμβάντων στην Ευρώπη. Τα δικαστήρια που ασχολούνται με τα θέματα αυτά χρειάζονται σαφείς ορισμούς. Η ιδέα ενός ευρωπαϊκού πλαισίου σημαίνει όχι μόνο ευαισθητοποίηση του κόσμου, αλλά και για την ποινική δίωξη μπορεί να είναι πολύ σημαντικό. Όλα ξεκινούν από έναν γενικό ορισμό της ανοχής. Είναι χρήσιμο λοιπόν να έχουμε ένα σαφές ε, πλαίσιο. Επικροτώ την προσπάθεια αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να επανέλθουμε στους προσκεκλημένους μας που θα κλείσουν τη συζήτηση αυτή. Να σας θυμίσω ότι καλέσαμε τους τρεις προσκεκλημένους μας να μας παρουσιάσουν την ε, πρόταση αυτή. ακολουθώντας ε, μια εντολή της διάσκεψης των Προέδρων. Χαιρόμαστε λοιπόν για τις παρεμβάσεις σας. Χαιρόμαστε που τονίζετε τη σημασία των αξιών και της δέσμευσης που απαιτείται ε, είναι πάρα πολύ σημαντικά τα θέματα αυτά για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Μπορείτε λοιπόν ε, να κάνετε μια δήλωση σχετικά με την κατάσταση που βλέπουμε όπου οι ιδρυτικές αξίες και αρχές που αποτελούν μέρος του ευρωπαϊκού DNA. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτές οι θεμελιώδεις αξίες ε, εξασθενούν. Και Ακόμα και εδώ μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βλέπουμε να συμβαίνει αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε. Σας έχουμε προσκαλέσει να παρευρεθείτε και με βάση τον κανονισμό. Ο καθένας μπορεί να πάρει το λόγο. Πρέπει να ομολογήσω ότι ντρέπομαι που δεν είχαμε περισσότερους βουλευτές σε αυτήν την σημαντική συζήτηση. Και λυπάμαι επίσης που αυτό έχει επηρεάσει την ε, ισορροπία στην αντιπροσώπευση των μελών. Κάποιες φωνές λοιπόν που θα έπρεπε να έχουν ακουστεί ήταν απούσες. Λυπάμαι γι' αυτό και ζητώ συγγνώμη στο όνομα της Επιτροπής. Σας δίνω το λόγο για να κλείσετε τη συζήτηση. Σας παρακαλώ να είστε σύντομοι διότι μας πιέζει ο χρόνος. Κύριε Τίνγκσταϊν κύριε Πρόεδρε. Ήθελα απλά να απαντήσω σε κάποιες τις παρατηρήσεις που έγιναν. Η πρώτη αφορά την ανοχή και τις διακρίσεις. Να σας θυμίσω ότι στη Σοβιετική Ένωση πριν την κατάρρευσή της, σε μια αθεϊστική χώρα ουσιαστικά υπήρχε μια θέση απέναντι στη θρησκεία που δεν είχε να κάνει με διακρίσεις, ήταν κατά όλων των ειδών ε, των θρησκειών, ε, κατά του Ιουδαϊνισμού, κατά του Χριστιανισμού. Ε, αυτό είναι διάκριση, όχι, είναι όμως μυσαλλοδοξία. είναι έλλειψη ανοχής και θα μπορούσα να σας δώσω πολλά άλλα παραδείγματα. Και είναι υποχρέωση της κυβέρνησης να εξαλείφει την μυσαλλοδοξία, όχι μόνο αυτήν καθ' αυτή, Ε, αλλά να λαμβάνει και όλα τα απαραίτητα βήματα στο πλαίσιο της δέουσας επιμέλεια, Όσον αφορά την εκπαίδευση, εγώ δεν είπα ότι πρέπει να διδάσκεται η ανοχή, αυτό δεν έχει νόημα. Θα πρέπει οι σπουδαστές να ε, αποκτούν επαφή με αυτό που θεωρούν ξένο και περίεργο, να καταλάβουν την, ε, την επικοινωμορφία. Δεν ε, είμαστε όλοι όμοιοι, δεν έχουμε το ίδιο χρώμα, δεν μιλάμε με τον ίδιο τρόπο, ούτε έχουμε όλη την ίδια θρησκεία. όσον αφορά την παρατήρηση που έγινε, την δίωξη ανθρώπων για τα όσα λένε, εκπλήσω κάθε συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λέει η ότι δεν επιτρέπεται να παρακινεί κανείς σε βίες πράξεις. Αυτό ε, είναι αδιαφυσβήτητο και στην Ρουάντα το Διεθνές Δικαστήριο ε, καταδίκασε ε, ανθρώπους για γενοκτονία για ομιλίες που είχαν κάνει. Ε, εάν πιστεύετε τέτοια πράγματα λοιπόν ζείτε σε άλλον κόσμο από μένα. Δεν πρόκειται για ε, ε, γνώμες ακαδημαϊκού επίπεδου. Είναι πράγματα σημαντικά και που αφορούν τον κόσμο στον οποίο ζούμε και θέλουμε να ζούμε. Εγώ δεν χρησιμοποίησα τον τον όρο προσελητισμό. Ο στόχος της εκπαίδευσης είναι να αποφευχθεί ε, ο προσελητισμός. Πρέπει να δείξουμε ότι υπάρχουν διάφορες απόψεις και ότι έχουμε δικαίωμα να είμαστε όλοι διαφορετικοί. Και όποιος πιστεύει ότι όλοι πρέπει να είμαστε οι ίδιοι ε, ε τι να σας πω... Ε, κύριε Ντίνσταϊν, σας ευχαριστούμε για τη δήλωση αυτή. Σας παρακαλώ να είσαστε σύντομος γιατί πρέπει να κλείσουμε. Μία πρόταση ακόμα. Ε, φυσικά είναι απαραίτητη η νομοθεσία. Εξίσου απαραίτητο είναι, και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που υπόθηκε, είναι ότι χρειάζεται ε, να υπάρχει δημόσιος διάλογος διαφανής ε, και ο κόσμος θα πρέπει να γνωρίζει τι διακυβεύεται. Και οι προτάσεις, οι, οι λύσεις δεν θα πρέπει να είναι αυτές που προτείνω εγώ, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν λύσεις. Κύριε Μπίλ, έχετε κάτι να προσθέσετε, κύριε Νέσιο, όχι. Εφόσον λοιπόν κλείσατε, σας ευχαριστούμε που ήσασταν ανάμεσά μας, ευχαριστούμε που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας και παρουσιάσατε τα επιχειρήματά σας για την προώθηση της ανοχής. Κάτι το οποίο θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό στην παρούσα φάση. Καλώς, θα ήθελα να περάσουμε λοιπόν τώρα στην ε, συνάντηση των συντονιστών. Ε, παρακαλώ αυτούς οι οποίοι δεν έχουν την, ε, την δυνατότητα ή το λόγο να πάρουν μέρος στην συνάντηση των συντονιστών να εγκαταλείψουν την αίθουσα. Μόνο όσοι έχουν την δυνατότητα να παραμείνουν.